Εάν θέλουμε να βάλουμε, που μπήκε σε νέε βάσεις τώρα το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, και θέλουμε να μπορούν να επιβληθούν και κυρώσει, πρέπει τότε να μην αμφισβητήσουμε αυτή την κοινή βάση. Έχεις δίκιο που λε ότι εάν το ερμηνεύσουμε με υπερβολικό τρόπο, τότε χάνουμε αυτή την ενιαία στέρη βάση όπου οι πολίτες ανεξαρτήτως χώρας, είτε από αυτές που έχουν μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες είτε όχι, οι ίδιοι αντιμετωπίζουν πια δυσκολίες. Και πιστεύω Γιάν, ότι μπορούμε, μπορείτε να καταλήξετε σε συμβιβασμό. Χωρίς να οδηγούμαστε διαρκώς σε υπονόμευση. Να πούμε ότι θέλουμε το Σύμφωνο σταθερότητα και Ανάπτυξης γιατί οφείλουμε να δώσουμε αυτή την ασφάλεια στους πολίτες την οποία τους χρωστάμε και οι οποίοι την περιμένουν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλος? Θέλει κανείς άλλο το λόγο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως? Όχι. Ωραία. Θα ψηφίσουμε αύριο. Και η Επιτροπή Περιφερειακή ανάπτυξη ελπίζουμε ότι θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μας. Θα ψηφίσει 11 και 12 Ιουλίου. Λέω θα λάβει υπόψη τη, αλλά δεν θα λάβει υπόψη τη αν ο εισηγητή δεν στηρίξει τη γνωμοδότησή του. Ξέρετε τι γίνεται. Αν η αν θέλουμε η γνωμοδότησή μας να λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια επί της ουσίας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, θα πρέπει να τη στηρίζουμε μέχρι το τέλος. Και το λέω αυτό γιατί συχνά με τις γνωμοδοτήσεις δεν ισχύει και είναι κρίμα. Να έχουμε επενδύσει τόση ενέργεια και τόσο κόπο και τελικά η θέση μας να μην λαμβάνεται υπόψη. Και ερχόμαστε στο σημείο 7 Εδώ θα εξετάσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες Πρώτοι για την έκθεση του κύριου Ταμάς Ντόιτς. Είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου όσον αφορά τον ε, κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και για τις διαδικασίες που αποσκοπούν στην διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών της Ένωσης στην αγορά τρίτων χωρών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Κάθε σχέδιο γνωμοδότησης που φτάνει στη δικιά μας Επιτροπή ασχολείται με πολύ σημαντικά ζητήματα. Και το κείμενο αυτό, του οποίου τον τίτλο διάβασε με απόλυτη ακρίβεια η Πρόεδρος, είναι σημαντικό. Θέλω λοιπόν εδώ να υπογραμμίσω ότι η γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής μας είναι η Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας, μιλάει για το εξή Πώς θα ανοίξουμε ή πώς θα διατηρήσουμε ανοιχτή την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις δημόσιες συμβάσεις τρίτων χωρών και πώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες. Ως συντάκτης της γνωμοδότησης αυτής θέλω πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω εδώ το θέμα της απασχόλησης. Και γι' αυτό θέλω αυτής εξ αρχής να ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές για το δικό τους έργο, που ήταν πραγματικά επικοδομητικό. Είχαμε 33 τροπολογίες εδώ στην Επιτροπή μας, πάνω στο κείμενο αυτό. Οι μισές αναφέρονται στο άρθρο 94 της Σύμβασης του Οργανισμού, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας που λέει ότι πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή 94 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, που όμως δεν έχει κυρωθεί ακόμα από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε από άλλες τρίτες χώρες. Και γι' αυτό ακριβώς σκέφτηκα ότι θα ήταν προτιμότερο να αναφέρομαι στην αιτιολογική σκέψη στη σύμβαση αυτή και όχι στα άρθρα. Με τους συντάκτες των τροπολογιών πάντως συμφωνήσαμε για το ότι αυτή τη λύση θα επιλέξουμε. Όσον αφορά τη Σύμβαση 94 της ε, ΔΟΕ. Υπάρχει μια τροπολογία βέβαια οριζόντια που την ακυρώνει και σε κάποιες άλλες τροπολογίες αναφερόμαστε στην διεθνή σύμβαση. Λέμε ότι είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Στο Στρασβούργο πάντως συνεδριάσαμε με τους κιόδες και μετά από τη συνάντηση αυτή διατυπώσαμε και 10 συμβιβαστικές τροπολογίες. Ένα μέρος αυτών είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα τροπολογίες και έχουν να κάνουν μόνο με αυτό, να μην συμπεριληφθεί δηλαδή στα άρθρα η μνήα στη σύμβαση αυτή της ΔΟΕ, αλλά να συμπεριληφθεί στην αιτιολογική σκέψη. Όσο για τις άλλες συμβαστικές τροπολογίες, αυτές καλύπτουν περίπου τις μισές από τις υπόλοιπες τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Όσες λοιπόν τροπολογίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβαστικέ, με εξαίρεση κάποιες πολύ λίγες, θα τις στηρίξω. Και μετά από την σημερινή μας συζήτηση θα καταλήξω και στον οριστικό κατάλογο ψηφοφοριών. Τώρα ποιες τροπολογίες δεν ε, θέλω. Είναι οι τροπολογίες 22 και 40. Σύμφωνα με τις δικές μου πεπιθήσεις, οι δύο αυτές τροπολογίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της γνωμοδότησης αυτής και γι' αυτό και δεν τη στηρίζω. Και άλλη μια φορά, ευχαριστώ πολύ όλους τους κοιόδες εισηγητές για τη βοήθειά τους και τις προτάσεις τους. Όπως επίσης και για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε. Περιμένω τις ερωτήσεις σας τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εσάς και τις και τους συναδέλφους και ζητώ συγγνώμη διότι μετά από την παρέμβασή μου είμαι υποχρεωμένη να εγκαταλείψω την αίθουσα διότι ψηφίζουμε στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών και πρέπει να σπέσω. Νομίζω ότι έχουμε κατορθώσει να συμφωνήσουμε επί συμβαστικών λύσεων πραγματικά εξαιρετικών με σαφείς κανόνες ό,τι αφορά την πρόσβαση υπηρεσιών και αγαθών στην ευρωπαϊκή αγορά αναθέσεων. Και αυτό είναι σημαντικό για μας ως Επιτροπή Απασχολήσεως. Είναι ένα μόνιμο θέμα, διότι πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζόμενων. Βεβαίως εκεί πρέπει να μπουν και πτυχές του περιβαλλοντικού δικαίου κλπ, διότι παραβιάσεις κατά των σχετικών κανόνων, εφόσον γίνονται διαρκώς και έχουν μια συγκεκριμένη βαρύτητα μπορούν να οδηγήσουν σε απαγόρευση μιας χώρας ε, από την πρόσβαση στις αγορές. Χαίρομαι που μπορέσαμε να συμφωνήσουμε επίσης ότι διεθνώς αναγνωρισμένες συμφωνίες πρέπει να περιληφθούν στην απόφαση αυτή. Η σύμβαση ILO της Διεθνούς Οργανώσης Εργασίας, δηλαδή 94, αναφέρεται στην έκθεσή μας. Εγώ θα ήθελα να αναφέρεται ακόμα πιο έντονα, αλλά και η συμβαστική λύση την οποία καταλήξαμε μας ικανοποιεί. Τονίζω ακόμη την τροπολογία 22, την οποία καταθέσαμε διότι επιθυμούμε να γίνει μια διασάφηση ότι αυτά που πράττουμε στο διεθνές εμπόριο δεν επιτρέπεται να οδηγήσουν στο να εξαναγκάσουμε τρίτες χώρες να ιδιωτικοποιήσουν την προσφορά υπηρεσιών τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο τονίσαμε κατ' επανάληψη και μέσα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων Παραχωρήσεων ότι οι χώρε μέλη είναι αυτέ που θα κρίνουν και θα αποφασίσουν αν θα ιδιωτικοποιήσουν ορισμένου τομεί ή όχι. Αυτή την ελευθερία αποφάσεω οφείλουν να την διατηρήσουν. Το ίδιο και για τι χώρε με τι οποίε συναλλασσόμεθα. Θεωρώ συνολικά ότι έχουμε μια στέρεα βάση για συζήτηση. Μπορέσαμε την προηγουμένη εβδομάδα να συμφωνήσουμε γρήγορα πάνω σε ορισμένα πράγματα και νομίζω ότι θα καταλήξουμε εύκολα σε μια κοινή θέση. Ευχαριστώ, Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Από την άποψή μου δεν υπάρχει ανακαιότητα να τεθεί θέμα κοινωνικών κριτηρίων για το εργαλείο πρόσβαση στην αγορά. Το λέω αυτό διότι αυτό περιλαμβάνεται επαρκώς στην οδηγία για τις επίσημες συμβάσεις αναθέσεων, όπου εγώ ως Γιώργης Συγητής συνδιαπραγματεύτηκα. Βεβαίως, για τις δημόσιες αναθέσεις αποδίδουμε σημασία στην δέσμευση των επιχειρήσεων στις προβλέψεις του νομοθέτη, να μην προχωρούν σε κοινωνικό ντάμπινγκ και άλλα σχετικά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μπει αυτό και εδώ. Πέραν αυτού, η εφαρμογή της οδηγίας δεν ανταποκρίνεται στη νομική βάση. Επαναλαμβάνω ότι εδώ πρόκειται μόνο για την αμοιβαιότητα, αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις αγορές αναθέσεων εκατέρωθεν. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να υποστηρίξω όλες τις συμβαστικές τροπολογίες. Για τις συμβαστικές α και β λένε ότι θεωρείται ότι λείπει η αμοιβαιότητα και όταν διακυβεύονται σημαντικά οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή η τήρηση σημαντικών περιβαλλοντικών κανόνων. Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες αναθέσεις τρίτων χωρών. Συμβαστική γάμα λέει ότι η Κομισιόν για την αξιολόγηση των σχετικών παραβιάσεων διερευνά το δίκαιο των τρίτων χωρών. Επίσης πρέπει να διερευνάτε κατά πόσον οι εκεί αρμόδιες αρχές για τις αναθέσεις κάνουν κοινωνικό dumping. Οι τρίτες χώρες δηλαδή αποκλείονται ή θα αποκλείονται συνολικά από τις αναθέσεις εάν έστω και μία επιχείρηση έχει παραβιάσει τις, ε, τους κανόνες αυτούς. Αυτό μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες ωστόσο για ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα πρέπει να διακρίνουμε εάν το κοινωνικό dumping γίνεται από επιχειρήσεις ή από αρχές. Η συμβαστική ΔΕΛΤΑ λέει αφενός πρέπει να γίνεται η συμβαστικη τα λεει αφενος εξέταση, δεύτερο για, τις, για τα, τα κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και αντί για τη χαμηλότερη τιμή το κριτήριο να είναι η βιωσιμότητα. Ίσως να δεχθώ εγώ το πρώτο, αλλά όχι εδώ στο άρθρο 6 που ορίζει τις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών για τον αποκλεισμό προσφορών από τρίτες χώρες. Σας μην λησμονούμε ότι πρόκειται για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας εδώ. Μετά έχουμε και το άρθρο 66 της οδηγίας περί συμβάσεων ε, αναθέσεων. Εδώ πέρα πρέπει να κρίνεται το οικονομικά, οικονομικά πλέον συμφέρουσα προσφορά. Όμως όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν ότι οι αναθέσεις θα γίνονται στη βάση της χαμηλότερης τιμής, εφόσον πρόκειται δηλαδή για τυποποιημένες υπηρεσίες ή προϊόντα. Έχουμε λοιπόν την ευκαμψία, έχουμε στο μέλλον την φθηνότερη τιμή και αυτό ρυθμίζεται βεβαίως στην οδηγία περί αναθέσεων. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιος άλλος να παρέμβει, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Oui, merci, Madame la Ευχαριστώ. Όπως υπενθύμησαν και πολλοί παρεμβαίνοντες, αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα ένας ε, τριμερής διάλογος για τη μεταρρύθμιση των οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες και γνωρίζετε ότι στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες γίνονται συζητήσεις και αναζητάται ένας συμβιβασμός. Όταν ασχοληθούμε με την εξωτερική πτυχή της ε, πολιτικής της εσωτερικής αγοράς, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχουν μια συνεκτική πολιτική. Κατανοείται λοιπόν ότι οι εργασίες αυτές είναι εργασίες αναφοράς για τη γενικότερη μας συλλογιστική, γιατί πολλοί από εσά ασχολείστε με το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή, να υπάρχουν κοινά σημεία αναφοράς με βάση τις ε, διαπραγματεύσεις ε, για την ε, αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επί τροπολογιών που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις υπό την μία ή την άλλη έννοια στις, ως προς τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, την έκβαση των οποίων δεν γνωρίζουμε ακόμα θα επανέλθουμε σε επιμέρους σημεία όταν χρειαστεί και όταν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Ο κύριος Ντόιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εντάχει και μόνο. Θα ήθελα να απαντήσω στον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κρίνουμε τη γνωμοδότηση, αλλά ίσως υπάρχουν και ορισμένες ε, αδυναμίες. Ε, ίσως δηλαδή εγώ δεν μπορώ να διευκρινίσω ορισμένα ζητήματα. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε προτάσεις συνδυασμού που ε, προβάλλουν εγγυήσει έτσι ώστε να μπορέσουν να υπερψηφίσουν οι περισσότεροι συνάδελφοι. Και όπως σας προείπα, οι τροπολογίες οι οποίες δεν καλύπτονται από τις τροπολογίες συμβιβασμού θα με απασχολήσουν. Θα έρθω σε επαφή με τους ε, συναδέλφους και θα καταρτήσω κατάλογο ψηφοφοριών αργότερα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας. Ευχαριστούμε πολύ, λέει και η Πρόεδρος, άρα θα ψηφίσουμε αύριο. Η Επιτροπή ΙΝΤΑ θα αποφανθεί το Νοέμβριο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουν ε, τα δικά μας, ε, τη δική μας συνεισφορά. Επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι το υπαριθμόν 8 και είναι... Ε, θα εξετάσουμε τις 12 τροπολογίες συμβασμού με βάση τις 144 που είχαν είναι οι δύο διασυνοριακές συλλογικέ διαπραγματεύσεις και ο διεθνικός κοινωνικός διάλογος. Ο κύριος Χέντελ, ο εισηγήτης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, 144 τροπολογίες. Και παρόλα αυτά, κατορθώσαμε, παρά το μεγάλο φάσμα που καλύπτουν οι τροπολογίες, κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε ορισμένες συμβαστικές τροπολογίες. Ακόμα βέβαια δεν είναι σαφές ποιες πολιτικές ομάδες και πώς θα τοποθετηθούν επ' αυτών. Μόλις χθες μπορέσαμε να διαβιβάσουμε τις ε, τροπολογίες, λυπούμε γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον από μια πολιτική ομάδα οφείλω να ε, τονίσω ε, προήλθαν πάρα πολλοί αποκλίνουσες τροπολογίες και γι' αυτόν τον λόγο ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβιβασμού. Ασφαλώς το θέμα είναι σημαντικό και χρειάζεται περισσότερη νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου. Κάτι που δεν είναι τόσο ικανοποιητικό είναι ότι σε όλες τις συζητήσει. όχι μόνο δεν λήφθηκαν υπόψη τα όσα συζητούνται γενικά στην Ευρώπη, αλλά δεν απορρίφθηκαν κιόλα. Ο κοινωνικός διάλογος δεν εξαρτάται μόνο από το ότι είναι ε, αναγκαίο από την άποψη της οικονομίας, αλλά ο διάλογος διεξάγεται επί ισότιμης βάσης. Αμφισβητείται λοιπόν η βάση, η δεσμευτικότητα είναι ανεπιθύμητη και μάλιστα αμφισβητείται ακόμη και το ότι την εντολή για τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν, να διαθέτουν τα εργατικά συνδικάτα και οι ε, οργανώσεις εργοδοτών. Οι τροπολογίες ενός συντονιστού μιας μεγάλης πολιτικής ομάδας θεώρησαν ορισμένοι ότι πρέπει να λυθούν ως βάση του κ. Όρη, οι τροπολογίες 87 και 105, αλλά στις συμβαστικές τροπολογίες πάλι ανετράπει αυτό. Για μένα δεν ήταν ξεκαθαρό. Δεν κατανοώ ορισμένε τροπολογίε. Ίσως βέβαια μπορέσουμε διμερώς να τι διευκρινίσουμε. τι τροπολογίε 106 και 99 του κ. Μπέκερ. Που τίνουν στην κατάργηση της δυνατότητας διαιτησίας. Και η τροπολογία 76 της κυρίας Κορνέλησεν που επιθυμεί την διαγραφή οποιασδήποτε εθελοντικής βάσης, ενώ υπάρχει πρακτική σε πολλές χώρες μέλη της εθελοντικής προσφυγής στην διατησία. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι έχει αποδείξει την αξία της η διαδικασία αυτή και δεν κατανοώ για ποιο λόγο ζητούν την απόρριψή της. Παρακαλώ λοιπόν να εξεταστούν οι συμβαστικές τροπολογίες πρώτα και να αποφασίσετε ποιος τις υποστηρίζει και ποιος όχι. Εγώ νομίζω ότι πολλές πολιτικές ομάδες καλύπτονται από τις τροπολογίες. Επίσης, δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε απόσταση από το επίπεδο της συζήτησης που διεξάγεται ούτως ή άλλως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Ο Όρι, η κυρία Κορνέλισεν. Καταρχήν ο κύριος ε, όρη Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Τόμας Χέντελ γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολο, δεν ήταν καθόλου εύκολες οι διαπραγματεύσεις που μας οδήγησαν μέχρι το σημείο αυτό και γνωρίζω ότι οι διαφορές ήταν πολύ μεγάλες και δεν ήταν καθόλου εύκολο να φτάσουμε σε τροπολογίες συμβιβασμού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ε, καλή ε, θέληση έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα σωστό ε, modus vivendi. Ε, δεν, πρόκειται, ε, δεν μόνο για συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συναντηθήκαμε και με τους συντονιστές και με τους σκιώδεις, αλλά και μέχρι αργά χτες άλλαξαν οι τροπολογίες συμβιβασμού. Ας τις δούμε λοιπόν μία προς μία. Η τροπολογία C αφορά μία διαγραφή και μπορούμε να τη δεχτούμε. Στην D δεν είχαμε πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα διότι βρίσκεται στο ύψος των προσδοκιών μας. Στην ε δεν μπορούμε να την δεχτούμε, αλλά δεχόμαστε την σίγμα ταφ. Ε, G δεν συμφωνούμε, H Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, αλλά μπορούμε να τη δεχτούμε. Άι, δεν συμφωνούμε. Και την, ως προς το απολογία επί της παραγράφου 11 μπορεί να γίνει αποδεκτή όπως ορίζεται τώρα. Με την L δεν συμφωνούμε. Με την τροπολογία συμβιβασμού M δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. I συμφωνούμε διότι ε, αναφέρεται στον αριθμό των ε, διεθνικών εταιρικών συμφωνιών, αλλά νομίζουμε ότι είναι υπερβολικός ε, η πρόοδος έχει επιτελεστεί. Μιλάμε για 244 ε, τέτοιες συμφωνίες, αλλά 15 εκατομμύρια εταιρείες, τέτοιες εταιρείες που είναι ε, ενεργές. Εάν πραγματικά ισχύει αυτή η τάση, ίσως θα πρέπει να την σχετικοποιήσουμε κάπως. Αλλά τα πράγματα κάπως διευκρινίζονται. Ε, ως προς την B, ίσως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη ότι δεν ανήκει σε αυτή την έκθεση, σε αυτό το σχέδιο. Έτσι βλέπουμε τα πράγματα Κορνέλισον και μετά Λούντβικσον. Ευχαριστώ. Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που έκαναν οι σκιώδεις, στις περισσότερες περιπτώσεις εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά. Παρόλο που δεν διαφωνώ για τη διάθεση επίτευξη συμφωνίας, παρόλα αυτά οι διαφορές είναι μεγάλες. Εμείς ως πράσινοι Είμαστε απογοητευμένοι επειδή διαπιστώνουμε ότι δεν είναι δυνατόν ως κοινοβούλιο για αυτήν την υπόθεση να τονίσουμε τον ισχυρό ρόλο των κοινωνικών εταίρων ε, στα πλαίσια της ε, δομής της οικονομικής διακυβέρνησης. Η συζήτηση αυτή πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να γίνει και μάλιστα τώρα, επειδή οι κοινωνικοί εταίροι και οι εργαζόμενοι μένουν πίσω στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων για την οικονομική διακυβέρνηση. Το μόνο λοιπόν που θα μπορούσα εδώ να κάνω είναι να ζητήσω από τις ομάδες να ξαναδούν τις τροπολογίες 62 και 63 που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί τον ισχυρό ρόλο των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνηση Ελπίζω να έχουμε μία έκθεση γενικά και θα προσπαθήσουμε να συμβιβαστούμε για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Θέλω να σχολιάσω μόνο επί της συμβαστικής 4 που λέει ότι, ότι οι κοινωνικοί εταίροι σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις Εδώ θα πρέπει να μιλάμε για την αυτονομία. Πρέπει να συζητήσουμε κατά πόση αυτονομία αυτή πρέπει να υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό εννοούν αυτοί οι οποίοι το υπέβαλαν. Δεν είναι πιο σημαντικό οι κοινωνικοί εταίροι να μιλούν για καλές συνθήκες εργασίας και τέτοια. Είναι ένα περίεργο κείμενο δηλαδή και ελπίζουμε να μπορέσει να τροποποιηθεί ώστε να ακούγεται πιο λογικό. Ευχαριστώ. Όλοι Λούπιτσον τώρα και μετά Ντύρχ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να αρχίσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε. Συζητήσαμε και είδαμε ότι πάμε όλοι προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Δύσκολο είναι να βρεθεί μια κοινή γραμμή. Εγώ μπορώ να καταλάβω και να συμφωνήσω με πολλές τροπολογίες, αλλά από την άλλη μεριά αυτές είναι δύσκολο να ενταχθούν στα πλαίσια της έκθεσης αυτής, χωρίς να αποκλίνουμε από την ουσία. Θα στηρίξω πάντως τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν, γιατί δεν μπορώ να καταψηφίσω τις επικρίσεις που γίνονται όσον αφορά τα κριτήρια για τις συλλογικέ συμβάσεις. Έτσι καλώς γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στην Επιτροπή και τις δύο πλευρές για την επίλυση διαφορών. Δεν θέλω να ξεχάσουμε το πού και πότε πρέπει να γίνονται διαπραγματεύσεις. Οι συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε μπροστά μας μπόρεσαν να επαναφέρουν κάποια ισορροπία. Διότι πρέπει να συμμετέχουν ε, βέβαια οι εργαζόμενοι, αλλά αυτό που δεν αναφέρεται με σαφήνεια είναι το πού και πότε θα συμμετέχουν. Σίγουρα υπάρχουν πολλές και διαφορετικές δομές. Τα συνδικάτα διαφέρουν μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά το βήμα πρέπει να γίνει. Προσβλέπω λοιπόν στην ψηφοφορία και ελπίζω οι συμβαστικές τροπολογίες να εγκριθούν. Ευχαριστώ. Άλλους, κανείς, μετά από την κυρία Χίρς, α, ο κύριος Κάσλερ, η κυρία Χίρς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ προς τον εισηγητή. Πρώτα γνωρίζω ότι η έκθεση δεν είναι διόλου απλή. Ευχαριστώ λοιπόν και για την διάθεση συνεργασίας και για το έργο που επιτελέσατε. Μαζί με τον Γιούργεν Κρόιτσμαν χειριστήκαμε το φάκελο αυτό και κάναμε και τη σχετική συζήτηση μέσα στα πλαίσια της ομάδας των φιλελευθέρων. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ως φιλελεύθεροι θεωρούμε πολύ σημαντικό τον κοινωνικό διάλογο και τους κοινωνικούς εταίρους θεωρούμε ότι είναι οι βασικοί φορείς οι οποίοι ε, μάλιστα ασκούν ε, θαυμάσια τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, νέες δομές, νέα γραφειοκρατία, η δημιουργία τέτοιων νέων δομών νομίζουμε ότι θα οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερα εμπόδια. Και αυτό δεν μπορούμε να το εγκρίνουμε, διότι ο κοινωνικός διάλογος είναι ανάγκη να διατηρεί κάποια ευκαμψία και να μην χωθεί σε ένα στενό κορσέ. Ευχαριστώ τώρα για τις συμβαστικές τροπολογίες, έστω και αν δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε όλες, ούτε θεωρούμε ότι έχουν καλύψει όλες μας τις ανησυχίες. Έρχομαι πιο συγκεκριμένα σε ορισμένα σημεία. επειδή είναι λίγες οι υπερεθνικές συμφωνίες, δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ειδικό ε, θεσμικό πλαίσιο. Νομίζω ότι αυτό προέκυψε και από τις συζητήσεις μας. Θα, συμφωνούσαμε όμως με την ιδέα να κάνει τη σχετική εξέταση η Κομισιόν. Βεβαίως ο συμβασμός υπερβαίνει το όριο αυτό και γι' αυτό δεν δεχόμαστε τη συμβαστική τροπολογία ε ως ομάδα των φιλελευθέρων. Μίλησα ήδη για την δημιουργία νέων διοικητικών δομών. Εμείς θεωρούμε ότι οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να αναζητήσουν και να εύρουν τον πιο ενδεδειγμένο δρόμο. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει νέα ευρωπαϊκή δικαιοδοσία. Και αναφέρομαι στις συμβαστικές τροπολογίες I και J, που όπως έχουν τώρα δεν μπορούμε να τις δεχθούμε. Κατά τα άλλα συμφωνώ με τον κύριο Όρη ότι η μακροοικονομικές ανισορροπίες κατά τη γνώμη μας δεν έχουν λόγο να περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Γι' αυτό και η συμβαστική Β ε, αντιμετωπίζεται κριτικά από εμάς, αλλά θα δεχθούμε τις D, H, καθώς και την Α. Ευχαριστούμε πολύ που ε, περιλάβατε το συγκεκριμένο νούμερο Θα εξετάσουμε επίσης τη συμβαστική τροπολογία γάμα, σε δηλαδή. Πολύ πιθανόν να την υποστηρίξουμε και αυτή. Έτσι λοιπόν εδώ τελειώνοντας επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου για την διάθεση συνεργασίας την οποία δείξατε. Ο κύριος Κάσλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Χέντελ, σε ευχαριστώ για την δουλειά που έκανες δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω με ορισμένα, έστω και αν διαπραγματευθήκατε συμβαστικές τροπολογίες και με τη δική μου πολιτική ομάδα. Εδώ τονίζω δύο πράγματα. Όλες μου οι τροπολογίες στρέφονται γύρω από την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Και θεωρώ ότι πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες χωρίς να δημιουργήσουμε νέο νομικό πλαίσιο. Εδώ υπάρχουν δύο λόγοι διότι αλλιώς βάζουμε τρικλοποδιά οι ίδιοι στους εαυτούς μας. Ούτε τα συνδικάτα, ούτε οι εργοδότες δεν συμφωνούν στις 27 χώρες μέλη. Δεν έχουν μια ενιαία άποψη δηλαδή για το πώς μπορούν να συναυθούν ευρωπαϊκές συλλογικές συμβάσεις. Ούτε επίσης θέλω να προκαταλάβω ένα ενδεχόμενο ευρωπαϊκό συντονισμό ενώ δεν γνωρίζουμε ποια κατεύθυνση θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο στενά θα διασυνδεθούμε ακόμη. Όχι λοιπόν νέες δικαιοδοσίες, ούτε δημιουργία νέων δικαιικών πλαισίων. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν σε ορισμένα με την συμβαστική γραμμή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για το άρθρο 74 δηλαδή τροπολογίες μάλλον, 71 και 84 διορθώνω, αυτές τις διατηρώ. Ευχαριστούμε. Άλλες παρεμβάσεις παρακαλώ. Όχι από ό,τι βλέπω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι. Κύριε Χάντελ, εσείς. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτα προς την κατεύθυνση της κυρίας περισσότερη γραφειοκρατία δεν προκύπτει ε, περισσότερη γραφειοκρατία αν υπάρξει μια ευρωπαϊκή ρύθμιση για την ε, ε, εθελοντική διαιτησία. Αυτό άλλωστε γίνεται σε υπερεθνικές συμφωνίες επιχειρήσεων. Δεύτερον, συμβαστική Β, εγώ την απέσυρα από τη βίστα ψηφοφορίας, δεν φάνηκε δυνατόν δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε συμβασμό στη βάση μονάχα μιας πολιτικής ομάδας. Το θέμα τέθηκε από τους πράσινους, το θέμα της μακροοικονομικής θεώρησης, που δεν είναι απαραίτητα δική μου ιδέα, αλλά ως στοιχείο περιλαμβάνεται στο κείμενο της εκθέσεως. Νομίζω εδώ θα χρειαστεί να ψηφίσουμε ξεχωριστά τις προτάσεις των πράσινων. Κάτι το οποίο βρίσκω ότι... Μάλλον ορισμένα από, τα, από, ορισμένες από αυτές με βρίσκουν σύμφωνο, ορισμένες όχι. Για τον κύριο Κέστλερ. Κάστλερ, συγγνώμη. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μιλούμε για ευρωπαϊκές συλλογικές συμβάσεις, ούτε την δημιουργία ευρωπαϊκών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κάθε άλλο. Εγώ θεωρώ ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν κανένα λόγο να ανακατευτούμε. Αυτό είναι καθαρά υπόθεση των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων. Ούτε είναι καν στόχος της εκθέση αυτής. Μιλούμε για συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων όπου υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας από τη μια μεριά ανάμεσα στις ηγεσίες των επιχειρήσεων και από την άλλη μεριά στα δικαιώματα των εργαζόμενων και στο τι προκύπτει ως διαφορά και πώς λύνονται οι διαφορές αυτές. Και όταν εξετάσουμε και ποιες θα είναι οι ανάγκες διαμεθοριακά της αναδιάρθρωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας, το πρόβλημα δεν είναι διόλου περιθωριακό. Θα έπρεπε προληπτικά να δημιουργήσουμε ένα εθελοντικό σύστημα που να επιτρέπει την εθελοντική πρόσβαση σε διαιτησία. Κύριε Κάστερ, δεν προχωρούμε δεν είναι στόχος μας δηλαδή να προχωρήσουμε σε, οποιοδήποτε συντονισμό μισθολογικό. Μιλάμε μονάχα για διαμεθοριακές συμφωνίες επιχειρήσεων, κυρίως για αναδιαρθρώσεις όπου υπάρχουν στο ευρωπαϊκό εκεί δικαιικό πλαίσιο ορισμένα κενά. Αυτά λέει η έκθεση. Το τι θα κάνει τελικά η Κομισιόν, υπάρχουν και σχετικά έγγραφα της ε, Κομισιόν και συνιστώ να τα μελετήσετε. Παρακαλώ η Επιτροπή και η Γραμματεία να με ή μάλλον οι πολιτικές ομάδες και η Γραμματεία άλλωστε να μου γνωρίσουν εγκαίρως ποιες συμβαστικές τροπολογίες υποστηρίζονται ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε και για την αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Ψηφίζουμε αύριο. Και το Σεπτέμβριο θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια. Ερχόμαστε στο σημείο 9. Πρόκειται για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την ευθύνη του κράτους σημαίας, της αρμοδιότητες του κράτους σημαίας. Είναι κάτι που σας έχω ήδη παρουσιάσει στις 30 Μαΐου, με λεπτομέρειες στις 30 Μαΐου του 2013. Τώρα απλώ θέλω να σας ενημερώσω για το ότι στην Κορεπέρ 12 Ιουνίου η Ιρλανδική Προεδρία επετέφθη συμφωνία επί του κειμένου αυτού. Έγινε μια τελευταία αναγκαία διόρθωση για τις επαρκείς δυνατότητες επιθεώρησης, κάτι το οποίο, μάλλον το Συμβούλιο δεν ήθελε να διευκρινίζουμε ότι έπρεπε να είναι επαρκής οι επιθεωρήσεις αυτές. Δεν νομίζω ότι βέβαια έχουμε κάνει συμφέρον να μπλοκάρουμε ολόκληρο το κείμενο, επειδή δεν δέχεται το Συμβούλιο αυτό το σημείο. Γι' αυτό και τελικά ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και ξέρω ότι η Ιρλανδική Προεδρία είναι ευτυχής που μπορεί να συμπεριλάβει το θέμα αυτό στον απολογισμό των δραστηριοτήτων της. Από κοινού με την έκθεση που είχε αναλάβει ο κύριος Μπράιαν Σίμψον στην Επιτροπή Μεταφορών για τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας στην Επιτροπή Μεταφορών εκείνος. Συνεπώς θα ψηφίσουμε αύριο τη συμβαστική αυτή πρόταση για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση που τον Οκτώβριο θα πάει στην Ολομέλεια εφόσον προηγουμένως οι ειδικοί γλωσσολόγοι νομικοί θα το έχουν ε, κοιτάξει πολύ καλά. Ο κύριος Σωρή. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά τη συμφωνία, πιστεύουμε και εμείς ότι είναι αποδεκτή και θα υπερψηφίσουμε αύριο. Αγαπητές και οδη εισηγητά από το ΕΛΚ, σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Όχι. Καλώς. Οπότε, ερχόμαστε τώρα στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Εδώ πρέπει να έχουμε μια κοινή συζήτηση για πρόταση προφορικής ερώτησης και πρότασης ψηφίσματος όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Στον τομέα αυτό, οι συντονιστές το ανέφεραν στην τελευταία συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο. Εδώ είναι τα σημεία 10 και 11 στην ημερήσια διάταξη και οι συντονιστές μου ζήτησαν να σας παρουσιάσω εγώ την κατάσταση. Έχει ως εξή. Θα θυμόσαστε ότι υπό την Καρίν Τελή στα μέσα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία που προβλέπεται για την περίοδο 2007-2012 είχαμε εγκρίνει έκθεση στην οποία ζητούσαμε η στρατηγική αυτή να ανανεωθεί. Τώρα έληξε, τελείωσε εδώ και 6 μήνες περίπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, καθυστερεί. Και δυσκολεύει την επεξεργασία του ζητήματος όπως θα έπρεπε. Οι συντονιστές λοιπόν εξέφρασαν την ανησυχία τους. Μάλιστα τώρα που βλέπουμε πως η κρίση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τους εργαζομένους και τους αναγκάζει να δέχονται συνθήκες εργασίες που κινδυνεύουν να τους εκθέσουν την υγεία τους και την ασφάλειά τους ακόμα περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν στους χώρους εργασίας. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι έπρεπε να στείλουμε ένα πολύ σύντομο μήνυμα στην Ολομέλεια, σαφές και αποτελεσματικό. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει η πρόταση για προφορική ερώτηση. Υπενθυμίζουμε πρώτα απ' όλα το πλαίσιο, το οποίο σας περιέγραψα κι εγώ, και απλώς ρωτάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συνέχεια θα δώσει σε αυτήν τη δημόσια διαβούλευση. Ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ή τέλο πάντων πολλοί από εμά καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να αποφύγει το ζήτημα. Οπότε ρωτάμε, ποια είναι τα εμπόδια το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνεχιστεί η στρατηγική αυτή. Να παρουσιάσει δηλαδή μια νέα τέτοια στρατηγική επιτροπή. Εμείς βέβαια τα ξέρουμε, αλλά πολύ θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας τα πει ρητά. Υπάρχει και ένα ψήφισμα, το οποίο υπενθυμίζει το νομικό και ιστορικό πλαίσιο που οδήγησε στην έγκριση της στρατηγικής αυτής και στη συνέχεια λέει ότι ανησυχεί και εκφράζει τη λύπη της που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άφησε να περάσει προθεσμία, ότι δεν προχώρησε και ότι το μήνυμα το οποίο είχε στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011. Το μήνυμα αυτό λοιπόν δεν εισακούστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά προτείνουμε. Σε όσου δεν συμμετέχουν στους συντονιστές τα λέω για να το ξέρετε και σας λέω επίσης ότι υπό αυτό το πνεύμα δούλεψαν και κατέληξαν σε αυτό οι συντονιστέ. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση επί της ουσίας, γιατί πιστεύουμε ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι κι αλλιώς έχει εκπονηθεί και έχουμε καταλήξει με το ψήφισμα αυτό του Δεκεμβρίου του 2011, άρα υπάρχει θέση του Κοινοβουλίου. Εδώ απλώς στέλνουμε ένα επιπλέον μήνυμα για να πούμε τι γίνεται. Ο κύριος Ευωρή και μετά ο κύριος Σέρκας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε, το μήνυμα αυτό, είναι ένα μήνυμα που μας βρίσκει σύμφωνος. Πάντα συμφωνούσαμε με αυτό. Το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία είναι δικιά μας αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Είναι ο τομέας ακριβώς όπου υπάρχει επίσης και ευρωπαϊκή κοινοτική αρμοδιότητα. Προβλέπεται σαφώς. Η νομοθεσία είναι δεσμευτική για όλες τις χώρες μέλη σε αυτό το τομέα. Άρα, η φόβοι, δεν ξέρω τι έκφραση ακριβώς να χρησιμοποιήσω, Πάντως το γεγονός ότι υπάρχει δισταγμός και δεν υπάρχει επιθυμία να ανανεωθεί η στρατηγική αυτή, ο φόβος αυτός που εκφράζεται όντως ισχύει. Και συμφωνώ με την Πρόεδρο ότι δεν πρέπει να ξανανοίξει η συζήτηση γιατί έχουν γίνει οι διαβουλεύσεις. Και δεν βλέπω πώς θα μπορούσαμε να είχαμε τροπολογίες σε μια τέτοια θέση. Εμείς μια γλωσσική τροπολογία μόνο έχουμε στείλει και πρόκειται για λεπτομέρειες. Συμφωνούμε επί της ουσίας. Ο Αλεχάνδρο Σέρκας και μετά η Τζιν Λάμπερτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς συμφωνούμε με την τοποθέτηση αυτή και εμείς έχουμε υποβάλει κάποιες μικρές τροπολογίες απλώς για να βάλουμε στο σημερινό πλαίσιο την ερώτηση και το ψήφισμα συμφωνώ και εγώ ότι επί της ουσίας έχουμε συμφωνήσει, δεν πρέπει να ξανανοίξει η συζήτηση. Έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα ουσίας, κυρία Πρόεδρο, όχι τόσο για τη στρατηγική, για την υγεία και για την ασφάλεια, αλλά για το τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γιατί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλήρως απούσα, όχι μόνο από αυτή την υπόθεση, αλλά και από άλλες υποθέσεις για τις οποίες θα έπρεπε να αναλαμβάνει πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπίσει και να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της, είτε πρόκειται για το πρωτογενές είτε για το παράγωγο δίκαιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ένα μόνο παράδειγμα από πολλά άλλα που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς για θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κοινωνικά, είτε για τους νέους είτε για οτιδήποτε άλλο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη στιγμή που είναι απούσα που δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία, από την άλλη μεριά προβάλλει ένα σωρό επιχειρήματα για να μην φέρει σε πέρα στις υποχρώσεις της. Ξεκινάει διαβουλεύσεις και ξανά διαβουλεύσεις. Μα έχει γίνει διαβούλευση, έχουν πει την απόψη τους όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Στο στάδιο που βρισκόμαστε δεν είναι δυνατόν να ανοίγει κι άλλη διαβούλευση μέσω ίντερνετ. πρόκειται για επιχειρήματα, όπως έγινε και με την αναδιάρθρωση. Καθαρά επιχειρήματα τα οποία εφεύρει για να μην προχωρήσει με την κοινωνική ατζέντα. Ενώ θα έπρεπε. Γι' αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή τις αρμοδιότητες της, τα καθήκοντά της. Είναι κατάλληλη στιγμή να το κάνουμε, κύριε Πρόεδρε. Τζιν Λάμπερτ και μετά Νάντια Χίρς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήμασταν ε, υπέρ του να θέσουμε το θέμα υπό τους όρους και αυτή ήταν και η αρχική πρόταση ε, για να δοθεί μια απάντηση. Αυτή θα είναι και η προσέγγιση όταν θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα. Όπως είπες, ήδη έχουμε ανταποκριθεί στην εργασία μας έτσι ε, ώστε να φτάσουμε και στα επόμενα στάδια της στρατηγικής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Θα πρέπει να δούμε πού είναι η στενοπή και πώς μπορούμε να τις υπερπούμε και αυτή την κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε στη διαπραγματεύση. Η Νάντια Χίρς. Και μετά θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα νομίζω το συζητήσαμε διεξοδικά και είναι και καλή έκθεση για τον τομέα της υγείας και της ασφάλειας από τους πράσινους. Ως Κοινοβούλιο λοιπόν έχουμε τοποθετηθεί. Και τώρα συμπληρώνεται το οπλοστάσιο με την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα. Και για την προφορική ερώτηση και για, την, ε, και για το ψήφισμα, τα κείμενα μας άρεσαν σε εμάς τους φιλελευθέρους, δεν θα κάνουμε λοιπόν, θα προτείνουμε άλλες αλλαγές, διότι νομίζω ότι οι διατυπώσεις οι δικές σας κύρια Πρόεδρε είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες και ως φιλελεύθεροι όπως είπα θεωρήσαμε ότι δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα που ενδεχόμενα θα αποδυνάμωνε το κείμενο. Όπως είναι λοιπόν τα σχέδια μας αρέσουν πολύ και τα υποστηρίζουμε ευχαρίστως. Euh, θα δώσω τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο, τον Βαϊτινό ε, ο οποίος θα μας εξηγήσει γιατί τέλος πάντων δεν εκπονείται αυτή η στρατηγική. Γιατί αργεί. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου, ε, η οποία ερχόταν από το Λουξεμβούργο, αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα στους σιδηροδρόμους και δεν μπόρεσε να προσέλθει. Θα είναι εδώ το απόγευμα για την ε, πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, της προτάσει για τους εργαζομένους η Επιτροπή δεν έχει και πολλά να πει, διότι, διότι γνωρίζουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Υπενθυμίσατε ότι η Επιτροπή συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για να δώσει τελική μορφή στη, στην προγενέστερη στρατηγική και μετά έχουμε προτείνει μία ανακοίνωση. Άκουσα το πολιτικό σας ε, ε, μήνυμα το δικό σας και των άλλων παρεμβενόντων. Θα ήθελα να σας πω ότι η απάντηση που ζητάτε ε, πάει πέραν από τις τεχνικές προδιαγραφές που θα μπορούσα εγώ να σας δώσω και θα σας απαντήσω ο ίδιος ο Επίτροπος στην Ολομέλεια. Ναι, λέει η Πρόεδρος και γι' αυτό προβάλλουμε αυτή την ε, προφορική ερώτηση με ψήφισμα στην Ολομέλεια Γι' αυτό την προτάσουμε γιατί είμαστε υπέρ των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στο διευθυντήριό σας. Ε, οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα αργές. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο την ε, προφορική ερώτηση και την πρόταση ψηφίσματος και θα ήθελα οι πολιτικές ομάδες να ασκήσουν πίεση στους συμμέτερους για να είμαστε όλοι παρόντες στην Ολομέλεια με την προφορική αυτή ερώτηση. Φτάνουμε λοιπόν... στο πιο θερμό σημείο τη σημερινής, του πρωινού μάλλον, που είναι το υπαριθμό 12. Τροπολογίες, θα εξετάσουμε τις τροπολογίες για τους αποσπασμένους ε, εργαζόμενους. Το σημείο αυτό προβλεπόταν στις 11. Θεωρώ ε, όμως ότι θα πρέπει να διακόψουμε λίγο γιατί η συγγήτρια δεν είναι παρούσα. Και ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς και από τους συναδέλφους πρέπει να διακόψουμε για ένα τέταρτο.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 Chers collègues, je vous propose de prendre... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, γιατί χρειαζόμαστε όλο το χρόνο μας. Είμαστε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Εξετάζουμε πρόταση συμβιβαστικών τροπολογιών σχετικά με την οδηγία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 96 κάθετος 71 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ μια ομάδα επισκεπτών που έχουμε. Είναι η κυρία Τσούβερ από το Υπουργείο Αποσχόλησης της Σερβίας. Και έχουμε και μία αντιπροσωπεία που τη συνοδεύει. Εκ μέρους όλων σας καλωσορίζω. Κυρία Χιασλοβιεύσκα, παρακαλώ, παρουσιάστε μας τις συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Από τον Φεβρουάριο, κάθε εβδομάδα Συνεδριάσαμε οι σκιώδες για να καταλήξουμε στις συμβαστικές αυτές τροπολογίες και εγώ ως εισηγήτρια ήμουν πολύ ανοιχτή στις προτάσεις όλων των πολιτικών ομάδων. Απόδειξη είναι ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αρχή πρόταση και τις συμβαστικές. Καταλήξαμε λοιπόν σε μια συμφωνία η οποία κατά τουλάχιστον 90% στηρίζεται από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες. Οι συμβαστικέ τροπολογίες, σύμφωνα με του κοινωνικού εταίρους, είναι λογικές, ισορροπημένε, κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο έργο, δεδομένου ότι αρχικά είχαμε 800 τροπολογίες. Δυστυχώ, βέβαια πρέπει να τονίσω ότι οι σοσιαλιστές όταν έκλειναν διαπραγματεύσεις τελευταία στιγμή πρότειναν τους δικούς τους συμβιβασμούς. Ακόμα και αν οι σοσιαλιστές ε, υπογράμμιζαν ότι δεν θέλουν συμβιβασμούς, τελικά οι προτάσεις τους βασίζονται σε αποφάσεις που είχαν ληφθεί νωρίτερα, αλλάζοντα που και που μια λέξη. Προσπάθησα να πετύχω συμφωνία μαζί τους, αλλά τελικά οι σοσιαλιστές αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις διαπραγματεύσεις. Από τα διάφορα άρθρα πρέπει να ξέρετε ότι είναι τα άρθρα 3, 9 και 12, εκείνα τα οποία είναι πιο επίμαχα. Το 3 έχει κατάλογο με διάφορα στοιχεία τα οποία θα εκτιμήσουν οι αρχές. Η πρώτη παράγραφος προβλέπει την υποχρέωση ελέγχου των ε, παράνομων αποσπάσεων. Οι εθνικές αρχές έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία και θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να επιλέγουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία παληθεύουν κάθε φορά. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχουν 27 χώρες από τις οποίες μόνο σε τρεις η απόσπαση γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Ο συμβασμός επί της παραγράφου 3 προτείνει να συμπεριλάβουμε και άλλα στοιχεία και περιλαμβάνει τα διάφορα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επαληθούν για να μην έχουμε ψεύδο Το άρθρο 9 τώρα αρχικά περιλάμβανε εθελοντική, εθελοντικά διάφορα στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι εργοδότες. Τα μέτρα ελέγχου προβλέπουν την κοινοποίηση, την υποχρέωση να υπάρχουν διαθέσιμα τα έγγραφα, η μετάφρασή τους, αλλά προβλέπεται και ο κατάλογος ατόμων επαφής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρέουν από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πολλές τροπολογίες έχουν προταθεί επί του άρθρου αυτού. Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αλλά καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που προβλέπει να ανοίξει ο κατάλογος ελεκτικών μέτρων και προβλέπει για τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν επιπλέον μέτρα και να ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τις άλλες χώρες μέλη. Τα μέσα αυτά πρέπει να αιτιολογούνται, δηλαδή πρέπει πράγματι να χρησιμεύουν για να αποφεύγονται οι καταχρήσεις και τα μέτρα να είναι ανάλογα με τον στόχο και όχι δυσανάλογα. Αν τον λέω θέλουμε να δούμε αν είναι νόμιμη μια εταιρεία ή όχι, δεν πρέπει να ρωτάμε το νούμερο παπούτσια φοράνε. Τρόπος του λέγει. Το σύστημα ελεγχού διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα της αγοράς εργασίας. Οι αρμόδιες αρχές λοιπόν έχουν την ελευθερία να επιλέγουν τα μέσα εκείνα τα οποία θεωρούν ότι είναι τα πιο αποτελεσματικά. Η υποχρέωση εφαρμογής και των τεσσάρων θα ήταν κάτι πολύ δεσμευτικό τόσο για τους εργοδότες όσο και για τον έλεγχο εργασίας. Οι ελεγκτές θα πρέπει τότε να αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο να ελέγξουν ένα σωρό έγγραφα σε ένα μόνο χώρο, κάτι το οποίο θα μειώσει την αποτελεσματικότητά τους για να καταπολεμήσουν την παράνομη απόσπαση. Ο συμβασμός για το άρθρο 12 επιτρέπει στις χώρες μέλη να υιοθετήσουν ένα αλληλέγγυο σύστημα βάσει των αρχών της μη διάκρισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίδια προστασία με τους τοπικούς εργαζόμενους. Μια τέτοια διάταξη διασφαλίζει ότι το σύστημα αλληλεγγύης δεν εφαρμόζεται μόνο στους αποσπασμένους εργαζόμενους. Τώρα έρχομαι στις συμβαστικές προτάσεις για την προστασία των εργαζομένων. Εκπονήθηκε από τους ε, σκιώδες εισηγητές και διασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της παροχής υπηρεσιών και την προστασία των εργαζομένων. Να κάποια παραδείγματα βελτίωσης τη κατάσταση όσον αφορά την απόσπαση. Πρόκειται για τον έλεγχο. Το άρθρο 3 περιλαμβάνει ένα κατάλογο στοιχείων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις ελεγκτικές αρχές να διαπιστώσουν αν μια επιχείρηση είναι απλώς με ταχυδρομική θηρίδα και τίποτα άλλο. Υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να εντοπίσουμε τι περιπτώσει αυτές των ψευδοανεξάρτητων. Το άρθρο 9 δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μέτρα επιπλέον ελέγχου ώστε να υπάρχει καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων που να προσαρμόζεται όμως τις διαδερότητες των χωρών μελών. Πρόσβαση τώρα στην κατάρτιση. Πού λέει επίμαχο θέμα. Ο συμβασμό επί του άρθρου 5 επιμένει στα δικαιώματα των εργαζομένων στην κατάρτιση. Όχι μόνο όσον αφορά τις ηθίκες εργασίας αλλά και την διαδικασία προσφυγής κατά των ε, μη έντιμων εργοδοτών. Μπορεί επίσης να υπάρξουν και σημεία επαφής. Οι εργοδότες πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει μετάφραση στην γλώσσα των εργαζομένων. Εγώ δεν καταλαβαίνω εδώ γιατί οι σοσιαλιστές ακυρώνουν τη δυνατότητα αυτή πρόσβασης στην πληροφόρηση με διαφάνεια. Γιατί δεν θέλουν να προβλέπεται αυτή η δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση και η ενημέρωση αυτή να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας ενώ από την άλλη μεριά παραδέχονται ότι υπάρχει ένα χάος στην ενημέρωση. Έπειτα έρχομαι στη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Ο συμβασμό για το σημείο 6 προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ανταλλαγή πληροφοριών χωρί καθυστέρηση όσον αφορά την απόσπαση. Κάθε άρνηση ενημέρωση από πλευρά των αρμοδίων αρχών καταγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιβάλλονται κυρώσει. Επίσης διατηρήσαμε την μικρή προθεσμία προκειμένου να μεταφέρονται οι πληροφορίες. Το άρθρο 8 τώρα επιμένει στο σύστημα IME, το οποίο προβλέπει ανταλλαγή γρήγορη και με ακρίβεια των πληροφοριών, προκειμένου να εμβαθύνουμε περισσότερο στη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών, κάτι το οποίο ζητούν και τα συνδικάτα. Το δικαίωμα τώρα προσφυγής. Έχουμε ένα σεβασμό στο άρθρο 11 που προβλέπει ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων κάθε φορά που θέλουν να προσφύγουν κατά των μη έντιμων εργοδοτών και διασφαλίζεται εδώ η νομική τους προστασία. Το ίδιο σκύει και για εργαζόμενους τρίτων χωρών. Επιπλέον προβλέπεται στο άρθρο 11 η υποχρέωση των κρατών μελών να δημιουργήσουν μηχανισμούς οι οποίοι να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να πάρουν το φιλόμενα. Και δεν βλέπω γιατί οι σοσιαλιστές εδώ προβλέπουν κάτι που δεν είναι αρκετά σαφές, ώστε τα συνδικάτα να μπορούν, χωρίς να ξέρουν καλά τους εργαζόμενους και την κατάσταση που επικρατεί, να ζητούν εκείνα τα οφειλόμενα. Δεν νομίζω ότι έτσι προστατεύουμε πραγματικά τους εργαζόμενους. Δεν ε, πετυχαίνουμε έτσι διαφάνεια. Έρχομαι τώρα στην αλληλεγγύη. Εδώ έχουμε μια συμβαστική πρόταση επί του άρθρου 12 που λέει ότι τα κράτη-μέλη τα οποία ε, αναλαμβάνουν το σύστημα αυτό αλληλεγγύης απέναντι στους αποσπασμένους εργαζόμενους να διασφαλίζουν την ίδια προστασία και στους τοπικούς εργαζόμενους. Η οδηγία για τους αποσπασμένους δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να προβλέψουμε μια τέτοια ευθύνη. Γνωρίζουμε από την πρακτική ότι δεν είναι ένα τέλειο μέσο η οδηγία αυτή. Δεν πετυχαίνει ο εργαζόμενος να πάρει το ποσό που του οφείλεται απλώς επιβάλλονται κυρώσεις στις χώρες. Εμείς με το συμβασμό εδώ προτείνουμε κάποιες διατάξεις που να είναι πιο αυστηρές σε εθνικό επίπεδο, που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των συνδικάτων και των εργαζομένων. Οι κυρώσεις τώρα. Τώρα τα 13-16 προβλέπουν απλούς κανόνες για την εφαρμογή των κυρώσεων διασυνοριακά τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τα ίδια κυρώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία για να διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες που δεν είναι έντιμοι τιμωρούνται. Σήμερα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μας χρειάζεται νομική σαφήνεια. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω όταν λέμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις στην περίπτωση που δύο οδηγίε δεν εφαρμόζονται στους αποσπασμένους, δεν καταλαβαίνω τη διατύπωση εδώ. Αν μας ενδιαφέρουν εδώ τα συνδικάτα, είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε με τους σοσιαλιστές, για τους οποίους η αρμόδια αρχή μπορεί να είναι και τα συνδικάτα. Πέρα δηλαδή από την επιθεώρηση εργασίας. Τα συνδικάτα δηλαδή θα μπορούν να έχουν όλες τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται και θα μπορούν να κάνουν ελέγχους, επιθεωρήσεις, να επιβάλλουν κυρώσεις και να ζητήσουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις κυρώσεις αυτές. Μα έτσι θα καταλήγαμε σε ένα γενικό χάος. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν παρά καμιά δεκαπενταριά επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν τον νόμο. Οι υπόλοιπε, που είναι πολύ περισσότερες, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Η υποχρέωση, η απέτηση μάλλον, αυτή για μας είναι παράδεκτη. Συχνά οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται για τις ανάγκες της απόσπασης. Η, τα γραφεία ενοικίασης εργαζομένων χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή. Εάν δεχτούμε τη διάταξη αυτή, αυτό σημαίνει ότι σε κράτη-μέλη όπως είναι η Γαλλία ή η Γερμανία, οι υπηρεσίες αυτές, τα γραφεία αυτά ενοικίασης εργαζόμενων δεν θα μπορούν να κάνουν αποσπάσεις. Για τα άτομα επαφή τώρα. Έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, η πρόταση των σοσιαλιστών προβλέπει υπερβολικά πολλά δικαιώματα. Το άτομο επαφής για τις συλλογικέ συμβάσεις θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα σε σχέση με το εμπορικό δίκαιο, για παράδειγμα. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ανθρώπους οι οποίοι δικαιούνται να κάνουν συλλογικές συμβάσεις. Εδώ αυτό που προτείνουν οι σοσιαλιστέ ξεπερνάει το ευρώ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πεδίο εφαρμογή αυτών των προτάσεων. Συνδικάτα και βελτίωση ηθικών εργασίας. Εδώ χαίρομαι πολύ γι' αυτό, ιδίως στη δικιά μου τη χώρα είναι στα συνδικάτα που οφείλουμε το 90% των βελτιώσεων. Οι δημόσιες αρχές όντως πρέπει να προχωρούν σε τέτοιες βελτιώσεις, αλλά πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα εκείνα που τους βοηθούν να είναι και οι κύριοι παράγοντες που θα προχωρήσουν σε αυτές τις βελτιώσεις και θα διευκολύνουν την σχέση ανάμεσα στην αγορά εργασίας και τους εργαζόμενους. Στο Συμβούλιο η κατάσταση ήταν δύσκολη, αλλά το Κοινοβούλιο πρέπει να θετήσει μια ισορροπημένη ε, πρόταση που να είναι αποδεκτή από όλους. Είμαι σίγουρη ότι ο συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε είναι εκείνος που μπορεί να βοηθήσει σε λύση. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ως πρόεδρος Επιτροπής να υπενθυμίσω έναν χρυσό κανόνα ε, λειτουργίας κατά τη διαπραγμάτευση μιας πρότασης νομοθετικού περιεχομένου. Όταν θέλουμε να φτάσουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, δεν θα ήταν σκόπιμο το Κοινοβούλιο να προτρέξει ως προς τη θέληση του Συμβουλίου. Εμείς είμαστε συνομοθέτες και ως από κοινού νομοθέτες θα πρέπει να προωθήσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου που εκλέγεται άμεσα από, πολίτες, από τους πολίτες για την περαιτέρω διαπραγμάτευση. Δεν μπορούμε να προτρέξουμε ε, ως προς τις επιθυμίες ορισμένων κρατών μελών ή του Συμβουλίου ε, γενικότερα. Αυτός είναι ένας ε, αναμφισβήτητος, αναμφισβήτητος κανόνας και μέσα στα πλαίσια του σε διαλόγου ξέρουμε όλοι πόσο ε, δύσκολο είναι να προωθήσουμε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Εμείς ε, ε, υποκείμεθα στη θέληση του Συμβουλίου, με συγχωρείτε που το υπενθυμίζω αυτό, αλλά επειδή μιλήσατε για μεθοδολογία στο τέλος της παρέμβασής σας, έκανα σκόπιμο να κάνω αυτή τη διασάφηση, να κάνω αυτή την διευκρίνηση, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να βλέπουμε και τη θέληση των κρατών. Εμείς δεν επιθυμούμε να ε, προβάλλουμε την θέληση των κρατών μελών. Ο Στίβεν Χιούζ. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ε, εισηγήτρια. Είμαι ευγνώμων για την εξαιρετική εργασία της εισηγήτριας εδώ και αρκετούς μήνες και για τους άλλους σκιώδεις. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ε, είπαμε ότι είμαστε δυσαρεστημένοι με την εξέλιξη των συζητήσεων, ιδιαίτερα ως προς τα άρθρα 3, 9 και 12. Λυπάμαι διότι δεν φτάσαμε σε συμφωνία ως προς το συνολικό πακέτο συμβιβασμών και χρειάστηκε να υποβάλουμε ξεχωριστές τροπολογίες, ιδιαίτερα ως προς τα τρία αυτά κρίσιμα άρθρα. Έχουμε αυτή τη σειρά των τροπολιών για την ε, ψηφοφορία αύριο. Προσπαθήσαμε να είμαστε απόλυτα σαφείς ορίζοντας τις προτάσεις μας σε σχέση με μια οδηγία ε, εφαρμογή που θα πρέπει να αποτελέσει συνέχεια της οδηγίας του 96 για τους αποσπασμένους ε, εργαζόμενους με βάση και τις υποθέσεις Λαβάλ ε, και Λουξεμβούρ που ε, εκδίκασε το ΔΕΚ και με βάση την απόφαση του ΔΕΚ. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία προσπαθήσαμε να έχουμε την περισσότερο δυνατή νομική ασφάλεια και θεωρούμε ότι θα, δεν θα υπάρχει τόσο υψηλή νομική ασφάλεια από ορισμένε προτάσεις της εισηγήτριας. Δηλαδή, μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση αντί να βελτιωθεί. Προτείνουμε ένα νέο άρθρο 1α για να συσχετίσουμε αυτή την οδηγία με το κοινοτικό δίκαιο και το κατεφαρμογήν δίκαιο. Επίσης, τι θεωρείται ε, θέμα δημόσια, δημόσιας αντιμετώπισης με βάση το άρθρο 3 σημείο 10, όπως αποφάνθηκε και το ΔΕΚ στην περίπτωση υπόθεσης του Λουξεμβούργου. Κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στο κείμενο της ε, εισηγήτριας. Στο άρθρο 11 ε, περιλαμβάνουμε το μοντέλο του Βόρα με μεγάλη σαφήνεια γιατί η απόφαση Λαβάλ ανέκυψε από υποθέσεις της Σκανδιναβίας. Και στο άρθρο 3 ορίζουμε ότι η πρόσληψη δεν πρέπει να έχει σκόπο απότερο σκοπό την απόσπαση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να διευκρινίσουμε την, να, να θέσουμε ένα πιο εύρωστο πλαίσιο για τη ε, νομική σαφήνεια και ασφάλεια. Για τα βασικά άρθρα 3, 9 και 12 νομίζω ότι το κείμενό μας είναι πιο σαφές. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει παράκαμψη και κατάχρηση της οδηγίας και θα πρέπει να δούμε πώς θα, αντιμετωπιστεί, θα αντιμετωπιστούν περιπτώσεις κατάχρησης. Έχουμε έναν ανοιχτό κατάλογο στο άρθρο 3 και στο κείμενο της εισηγήτριας καθώς και στο συμβασμού υπάρχει ένας ανοιχτός κατάλογος αλλά στη νέα στις νέες παραγράφους του άρθρου 3 αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέψουν επιπρόσθετους όρους τη στιγμή που είναι αιτιολογημένα αναλογικά και δεν προβαίνουν σε διακρίσεις. Όμως υπάρχουν δυσκολίες, γιατί ποιος θα αποφασίσει τι είναι αιτιολογημένο και αναλογικό. Ε, υπάρχει μεγαλύτερη ε, νομική ανασφάλεια και ανοίγει ορισμένες δυνατότητες. Δηλαδή έχουμε έναν ανοιχτό κατάλογο αλλά μπορεί να κλείσει. Στην ε, υπόθεση Viking θυμόσαστε πολύ καλά πόσο ε, τη στενή ερμηνεία, συσταλτική ερμηνεία είχαμε της αναλογικότητας. Σε αυτή την υποπαράγραφο η εισηγήτρια τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό σε μία ενιαία ιστοσελίδα. Αυτό το συζητήσαμε στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως σε έναν ιδεώδη κόσμο θα μπορούσαμε να είχαμε μία ενιαία εθνική ιστοσελίδα υποβολής. Αλλά είμαστε αρκετά μακριά και δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος ε, δυνατός τρόπος δεν ξέρω πόσο σε ένα ομοσπονδιακό κράτος θα μπορούσε να λειτουργήσει μία ενιαία ιστοσελίδα. Στο άρθρο 9 για τα εθνικά μέτρα ελέγχου έχουμε το πυρήνα των εθνικών επιθεωρήσεων και τα άλλα θέματα ε, απόκεινται στη διακριτική, εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Δεν ξέραμε αν πρέπει να βάλουμε ένα σαλ ή στο άρθρο 9. Έχουμε λοιπόν έναν πυρήνα και μετά το στοιχείο της διακριτικής ευχέρειας ε, στο ε, άρθρο 12 για την υπεργολαβία. Με την τροπολογία μας ορίζουμε την ευθύνη των ε, υπεργολάβων. Πρόκειται για ένα πιο λακωνικό κείμενο που ελπίζω να υποστηρίξετε. συνεργαστήκαμε και με το ETUC, με, την εθνική μας ε, συνομοσπονδία και με την FIC ε, από τον τομέα ε, των κατασκευών, έτσι ώστε να φτάσουμε σε τροπολογίες συμβιβασμού για τα άρθρα 3 και 9. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω στο Δινεκές. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα θέμα που έθιξε ο Σάμπα Όρη την τελευταία φορά. Ε, μιλήσαμε για έγκαιρη προειδοποίηση ε, σε σχέση με τους αποσπασμένους και μας είπε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων εγγυήσεων που θα πρέπει να ε, διασφαλιστούν σε περίπτωση απόσπασης. Θεωρώ ότι στην αρχική οδηγία στο άρθρο 3.2 Υπάρχει μία εξαίρεση για αυτό το συγκεκριμένο σημείο ε, έτσι ώστε να υπάρξει εγγύηση εργασίας για οκτώ ημέρες ε, τουλάχιστον μέσα στα πλαίσια της απόσπασης. Θα παραμείνω εδώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Η Νάντια Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα, θερμές ευχαριστίες προς την εισηγήτρια διεξήχθησαν πολλές και μακρές και πλούσιες σε χαρτί, αν μπορώ να το πω έτσι, συνεδριάσεις. Πραγματικά ήταν μεγάλο το έργο που αναλάβαμε και νομίζω ότι της αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ και έπαινος για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε την εργασία. Από την αρχή είχαμε μεγάλη απόσταση Βέβαια γνωρίζαμε ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια προσεγγίσεως για να συντάξουμε γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρήκα την εισηγήτρια να διαθέτει μεγάλη διάθεση συνεργασίας, να μετακινηθεί και από την θέση της και εμείς βεβαίως οι φιλελεύθεροι μετακινηθήκαμε από τις δικές, από τις δικές μας σε ορισμένα άρθρα εμείς είχαμε βάλει κάποιες κόκκινες γραμμές οι οποίες σιγά σιγά μεταχρωματίστηκαν σε χρώμα πορτοκαλί και κίτρινο, δηλαδή έγιναν λιγότερο απόλυτες και αυτό είναι το νόημα βέβαια του συμβιβασμού. Καταλήγουμε τώρα σε δύο διαφορετικές συμβιβαστικές γραμμές που καλούμεθα να ψηφίσουμε της συγκεκριτρίας και των σοσιαλδημοκρατών. πρώτη φορά για μένα αυτό. Βέβαια, ίσως έχει ξανασυμβεί αλλά πάντως νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχής ο τρόπος αυτός να ε, προβάλλονται, να, να κατατίθενται δηλαδή και εναλλακτικέ επιλογές. Νομίζω πάντως ότι μπορούμε αύριο να διεξαγάγουμε μια αρκετά λογική ψηφοφορία. Προσωπικά και για την ομάδα των φιλελευθέρων μπορώ να πω ότι για μας είναι σημαντικό να μην χάσουμε από τα μάτια μας την ευρωπαϊκή αγορά. Να μην προωθήσουμε τα προστατευτικά μέτρα. Πολλές από τις συμβαστικές ε, προτάσεις των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα τις εξετάσουμε. Εσείς είπατε ότι χρειάζεται ασφάλεια δικαίου. Υπάρχουν ωστόσο μέσα, περιλαμβάνονται μέσα πολλές προστατευτικές διαστάσεις, τις οποίες εμείς θέλουμε να αποτρέψουμε ωστόσο. Γι' αυτό δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις συμβαστικές προτάσεις των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών μίλησε κάποιος για την ιστοσελίδα. Από την αρχή τέθηκε το θέμα αυτό. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζονται πληροφορίες, ορθές πληροφορίες. Γι' αυτό λέμε ότι να υπάρχει μια μοναχή ιστοσελίδα. Οι χώρες μέλη μπορούν να εκδώσουν και φυλάδια αν θέλουν, αλλά να υπάρχει ένα homepage όπου να μπορεί να βρει κανείς τις απαραίτητες πληροφορίες. Ένα άλλο που είναι σημαντικό και περιλήφθηκε σε διάφορα άρθρα, διότι είναι κυρίως η προστασία του εργαζόμενου και για να προστατευτεί πρέπει να γνωρίζει τι περιλαμβάνει η σύμβασή του. Και για ελέγχου βεβαίως και τα σχετικά είναι απαραίτητο, να μπορεί να γνωρίζει κανείς περί τίνο πρόκειται. Γι' αυτό και επιμείναμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ευρύ φάσμα γλωσσών. Βεβαίως τα αγγλικά θα χρησιμοποιούνται καταρχήν εφόσον κινούμεθα προς την κατεύθυνση μιας ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό θα πρέπει, σε αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούν βεβαίως και οι αρχές. Στο άρθρο 9 δεν χρειάζεται να σας κρύψω ότι εμείς ήμασταν υπέρ της κοινοποίησης, notification. Δεχθήκαμε εν τέλει το inform in advance που είναι βεβαίως πολύ αποδυναμωμένο. Ίσια, ίσια μπορούμε να το δεχθούμε εμείς ως φιλελεύθεροι. Θεωρούμε όμως και εδώ ότι χρειάζεται αυτό το ανοιχτό πνεύμα Εάν τροποποιηθεί και αυτό, τότε νομίζουμε ότι υπερβαίνουμε το στόχο και μπαίνουμε πλέον σε ένα προστατευτικό πνεύμα το οποίο εμείς οι φιλελεύθεροι απορρίπτουμε. Στην παράγραφο 12 νομίζω κατέληξε σε καλή συμβαστική λύση η εισηγήτρια. Οι χώρες μέλη μπορούν να διατηρήσουν το σύστημα το οποίο διαθέτουν, επομένως η γενική ευθύνη παραμένει όπου υπάρχει Μπορούν, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες να το διατηρήσουν. Εμείς ωστόσο ξεκαθαρίσαμε τους στόχους ότι δηλαδή οι εργαζόμενοι λαμβάνουν το μισθό τους, καταβάλουν κρατήσεις για τις εθνικές ασφάλειες, είναι καθαρή στόχη λοιπόν. Πώς θα το ρυθμίσουν οι χώρες μέλη είναι δική τους υπόθεση και νομίζω και εδώ είναι ορθός ο συμβιβασμός. Συνολικά νομίζω, με, θεωρούμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε τις συμβαστικές λύσεις της εισηγητρίας και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αύριο με την ψηφοφορία, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο που και αυτές δεν διαγράφονται πολύ απλές και εύκολες. Καλά θα ήταν λοιπόν να υπάρξει μια ξεκάθαρη γραμμή αύριο της Επιτροπής Απασχολήσεως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ευθέω πλέον, ευθύ αμέσως πλέον στη διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Σρέντερ και μετά το Μασχάντελ. Αγαπητοί συνάδελφοι όμως, κάνατε μια παρατήρηση για την παρουσίαση των συμβαστικών προτάσεων. Θέλω απλώς να σας υπενθυμίσω στην προηγούμενη ψηφοφορία τη σημαντική που είχαμε στην Επιτροπή μας, εσείς οι ίδιοι με την ομάδα σας συνεισφέρατε στο να υποβληθούν συμβιβαστικές τροπολογίες εναλλακτικέ για όλες τις ψηφοφορίες για τις οποίες η εισηγήτρια είχε υποβάλει συμβαστικές τροπολογίες. Ήταν η έκθεση MR Costello, έτσι, για το Ταμείο πόρων. Συνεπώς, να κοιτάξει ο καθένας να δει τι κάνει ο ίδιος και ας προσπαθήσουμε να είμαστε επικοδομητικοί. Γιατί δεν μας εκπλήσει που υπάρχουν θέσεις στις οποίες μένει κανείς μέχρι το τέλος. Είμαστε εδώ για να τις συζητάμε. Η κυρία Σρέντερ πρώτα και μετά κύριο κύριος Ευχαριστώ. Η τελευταία σας παρατήρηση μου υπενθυμίζει ότι θα ήθελα να πω ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν πραγματικά επικοδομητικές, πραγματικά επικοδομητικές, επαναλαμβάνω, από την πλευρά της εισηγητρίας, η οποία φάνηκε ανα πάσα στιγμή διατεθειμένη να μετακινηθεί και υπέρ των υπολείπων. Καταλήξαμε σε κοινού συμβιβασμούς μέχρι την τελευταία συνεδρίαση. Τα πιο δύσκολα, οι πιο δύσκολες παράγραφοι ήταν 3, 9 και 12, όπου μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση. Και όλοι όσοι παρέστησαν στις διαπραγματεύσεις και μέχρι τώρα ήταν διατεθειμένοι ή διατεθειμένες να καταλήξουν σε αυτούς τους συμβασμούς. Βέβαια, δεν κατέστη αυτό δυνατόν, διότι Εν τέλει κατατέθηκαν εναλλακτικέ συμβαστικέ τροπολογίε, τι οποίε δεν είχαν διαπραγματευτεί οι καταθέτοντε με κανέναν. και που χαρακτηρίστηκαν και αδιαπραγμάτευτες. Η δυνατότητα δηλαδή που είχαμε προτείνει εμείς οι πράσινοι να πούμε το ένα σύνολο, ε, το ένα σύνολο συμβιβασμών μαζί και με το άλλο να τεθούν ξανά υπό διαπραγμάτευση για να καταλήξουμε σε μία ενιαία συμβαστική λύση, η αυτή δεν ήταν δεδομένη, ώστε να έχουμε ένα σύμβασμο ανά άρθρο. Αυτό θέλουμε εμείς. Το γεγονό ότι δεν κατέστη δυνατόν αυτό, οδήγησε εμάς τους πρασίνους να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση. Εν προκειμένου, λάβαμε λοιπόν τη δική μας γραμμή, είχαμε τη δική μας πράσινη εκδοχή, την οποία θεωρήσαμε ως δική μας κατευθυντήρια γραμμή. Αυτή η πράσινη εκδοχή ήταν η καθοριστική γραμμή για μας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις διάφορες συμβαστικές προτάσεις. Στόχος μας ήταν να συντάξουμε μια νομοθεσία η οποία να είναι πραγματικά στεγανή αποτελεσματική και η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί πραγματικά στην πράξη. Έχουμε το γεγονό ότι έχουμε μια ανοιχτή ενιαία αγορά και η νομοθεσία ως στόχο πρέπει να έχει να θεσπίζει καθαρούς κανόνες για την ενιαία αγορά και σε αυτούς συγκαταλέγεται ασφαλώς και ανάγκη βελτίωσης της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια αυτής της αγοράς. Αυτό για μας ήταν κεντρικό θέμα. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι σαφές ότι είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών, όπως άλλωστε το προβλέπει η υφιστάμενη οδηγία. Αυτές καθορίζουν και ελέγχουν τους ελάχιστους κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Ο έλεγχος αυτός είναι σημαντικό να μπορεί να διεξάγεται ελευθέρως, διότι η πράξη έδειξε ότι εάν δεν μπορεί να γίνει προσαρμογή στην κατάσταση, ο έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός και αυτό αποβαίνει εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και της προστασίας των ασθενέστερων σε αυτή την υπόθεση της απόσπασης εργαζόμενων. Και γι' αυτό θεωρήσαμε και εμείς ότι στο άρθρο 3 πρέπει να υπάρχει επαρκές περιθώριο ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή στην εκάστοτε διαμορφούμενη κατάσταση. Και τότε μόνον θα είναι δυνατόν να είναι αποτελεσματική η σχετική νομοθεσία. Εμείς δηλαδή ήμασταν απολύτως αντίθετες με την οδηγία εφαρμογής η οποία να τροποποιεί την αρχική και να υπάρχει τροποποίηση της κατανομής των αρμοδιοτήτων που προβλέπεται ούτως ή άλλως στην συνθήκη όπου οι κανόνες του δικαίου είναι αρμόδια, είναι αρμόδιες, για αυτές είναι αρμόδιες οι χώρες και ξαφνικά να γίνει αρμόδια η Κομισιόν. Και οι δύο μορφές των διαφόρων συμβαστικών τροπολογιών εξετάστηκαν από εμά λέξη προς λέξη, καθώς επίσης και οι σχετικές τους συνέπειες για την ομοθεσία. Και σύμφωνα με αυτή τη μελέτη θα ρυθμίσουμε την στάση μας στην ψηφοφορία και βάσει αυτής αποφασίσαμε ποιες τροπολογίες θα υποστηρίξουμε. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο κινήσεως και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε διότι ειδικά σε αυτά τα δύσκολα άρθρα όπως το 9 έχουμε αφενός την κατάσταση ότι χρειαζόμαστε ανοιχτό κατάλογο χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, γιατί μπορεί να τύχει ωστόσο η δεσμευτικότητα να οδηγήσει σε κλειστό κατάλογο. Εγώ έχω άλλη άποψη εδώ από τον Στίβεν Hughes, ότι αυτό δεν, είναι σωστό, δεν θα ήταν σωστό στην περίπτωση αυτή. του άρθρο 9 βέβαια έχει άμεσα σχέση με το γεγονός πώς γίνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κομισιών και χώρων μελών και εάν το άρθρο 5 της αρχικής οδηγίας θα παραμείνει ενισχύ ή όχι. Αυτό δε προκύπτει από μια λεξούλα στην διατύπωση της συμβαστικής τροπολογίας της Ντανούτα. Αυτό που ζητούν οι φιλελεύθεροι, δηλαδή αυτό το in advance, εκ των προτέρων. Αυτή τη στιγμή ισχύσει αυτό το in advance και όχι η κοινοποίηση προς την Κομισιόν, ώστε και οι άλλες χώρες να μαθαίνουν τι συμβαίνει ε, στις ε, υπόλοιπες, να υπάρχει ροή των πληροφοριών και το άρθρο 4 βεβαίως, που για μας έχει ιδιαίτερη σκοπιμότητα. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση άλλωστε της Ντανούτα και το υποστηρίζω εγώ, αλλά από τη στιγμή που μπαίνει το in advance προκαλούμε μια νομικά περίπλοκη κατάσταση διότι είναι διόλου καθαρό πλέον εάν μια χώρα μέλος οφείλει να αντιδρά με ελέγχους ή αν μπορεί. Και εκεί λοιπόν ανοίγουμε παραθυράκια. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τις αγγλικές λέξεις without delay, χωρίς καθυστέρηση, που προκύπτει και από το νόημα της, ε, του αρχικού άρθρου 4 και μπορεί να λειτουργήσει, διότι έτσι υποχρεούνται οι χώρες μέλη να κοινοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε οι άλλες χώρες μέλη να μπορούν να πληροφορούνται περί τίνος πρόκειται. Και η Κομισιόν τότε παίζει ένα σημαντικό συντονιστικό ρόλο και πρέπει να τον παίξει. Όμως, άλλος ρόλος της Κομισιόν στο θέμα αυτό δεν έχει νόημα. Αυτό για μένα είναι κεντρικό θέμα, διότι εν προκειμένου θα είναι κρίσιμο για μας για να αποφασίσουμε πώς θα ψηφίσουμε στο τέλος. Αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και μακρηγόρησα λίγο περισσότερο για να εξηγήσω ότι αυτό για μας είναι κέριο θέμα. Το άρθρο 3, όπως το διαπραγματευτήκαμε με την εισηγήτρια, Θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντικό και προτιμότερο διότι είναι συνεκτικότερο και στην ουσία καλύτερη νομοθετική ρύθμιση από την εναλλακτική επιλογή που προτείνεται και γι' αυτό το προτιμούμε διότι η εναλλακτική επιλογή που προτείνεται έχει σημαντικές νομικές ελλείψεις. Για το άλλο 12 το θέμα που τίθεται για μας τους πρασίνους είναι πολιτικό και είναι σαφές και το τονίζω επίσης εδώ, ότι στη διαπραγμάτευση υπήρξε πραγματικά πολλή κίνηση. Μετακινήθηκε σημαντικά η εισηγήτρια. Βέβαια, εάν τώρα πρέπει να κρίνω πολιτικά ποια είναι η προτιμότερη νομοθετική ρύθμιση, τότε για μένα είναι καλύτερα να μην είμαι υποχρεωμένη να μένω στο πρώτο στάδιο της γενικής ευθύνης, αλλά σε όλα τα στάδια από εκεί θα εξαρτηθεί η δική μας στάση στο θέμα αυτό. Παρόλο που τονίζω και πάλι ότι η πρόταση της ηγητρίας είναι καλύτερη, άλλωστε την διαπραγματευθήκαμε μαζί, καλύτερη από την πρόταση της Κομισιόν. Σαφώς καλύτερη. Και αυτό θα επηρεάσει βεβαίως την στάση μας στην ψηφοφορία. Αυτά για τα γενικά. Πιστεύω ότι θα είναι χαόδης η ψηφοφορία αύριο και είναι κρίμα. Τονίζω όμως και πάλι ότι ασφαλώς αυτό δεν βαρύνει την εισηγήτρια, η οποία έπραξε πάντα το δυνατό για να καταλήξουμε σε μια καλή ψηφοφορία. Τόμας Χέντελ. Τέτοιες οδηγίες γίνονται μόνο για να ενισχυθούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Επομένως, αυτό το δόγμα ότι δήθεν δεν πρέπει η νέα οδηγία να είναι καλύτερη από την προηγούμενη είναι εντελώς εσφαλμένο. Και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων είναι για μας ανεπαρκή. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, γι' αυτό θα περιοριστώ σε τρία σχόλια. Πρώτα, παράγραφος 3 αυτά που έχουν σχέση με το Ρώμα 1 και αν θα προβλέπετε ότι στην χώρα υποδοχής εφαρμόζονται οι σχετικές συνθήκες διότι δεν περιλαμβάνονται εδώ οι συλλογικές συμβάσεις. Επομένως, οι προτάσεις που έχουν γίνει εδώ είναι ανεπαρκείς και ιδίως εφόσον το βάρος της αποδείξεως φέρει ο εργαζόμενος. Στην πράξη διαπιστώνουμε συχνά ότι ο εργαζόμενος και λόγω της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και της επαπειλούμενης νέας κατάστασης δεν είναι σε θέση να προσφέρει, δεν είναι σε θέση να αναλάβει το βάρος της αποδείξεως. Για το άρθρο 9, εμείς ήμασταν από την αρχή κατά της κοινοποίηση. Αυτό φαίνεται πως έχει τροποποιηθεί μένα αλλά για μας ανεπαρκώς. Εμείς προτιμούμε ανοιχτή λίστα, ανοιχτό κατάλογο. Άνευ όρων, διότι μόνο έτσι θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Και οι χώρες μέλη το ίδιο, διότι ως Ευρωπαίος νομοθέτης γνωρίζουμε ότι μπορεί εμείς να δουλεύουμε πάνω σε μια νέα νομοθετική ρύθμιση, αλλά όποιες στρατιές από think tank ψάχνουν να βρουν άλλες δυνατότητες. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε εμεί ότι οι μηχανισμοί ελέγχου θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι και θα μπορούν να προσαρμόζονται. Ορισμένες νομικέ έννοιες όπως ενδεδειγμένο ή ανευθιακρίσεων κλπ. μου φαίνονται εντελώ ανεπαρκείς. Τέλος, γενική ευθύνη των επιχειρήσεων. Αυτό εμείς πρέπει να αποφύγουμε εδώ, πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε αποδυνάμωση και για τους περαιτέρω υπεργολάβους. Δεν μου αρκούν τα προβλεπόμενα για την ώρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει καθαρά να ενισχύσουμε και όχι να αφήσουμε σε μια φαιά ζώνη την μελλοντική εξέλιξη. Η μέχρι τώρα γενική, συνολική ευθύνη των επιχειρήσεων που ε, υφίσταται τώρα πρέπει να διαφυλαχθεί. Οι συμβαστικές τροπολογίες των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών μας βρίσκουν περισσότερο σύμφωνους από τις τροπολογίες της Συγγήτριας. Γι' αυτό και θα τις υπερψηφίσουμε αύριο. Τώρα μια τελευταία παρατήρηση στην διαβίβαση των τροπολογιών χάθηκε ένα δικό μας άρθρο. Η γραμματεία βέβαια μετά από συνεννόηση μαζί μας θα το περιλάβει. Νομίζω ότι θα είναι το μη μη 3 στο άρθρο 12. Εμείς το υποβάλαμε εμπροθέσμος. Αλλά μπορεί να συμβούν τα πράγματα αυτά, δεν με κανένα. Είναι όμως σημαντικό ε, να μνημονευτεί ότι πρέπει να περιμένετε κάτι της ακόμα από μας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Τώρα θα λάβουν το λόγο οι άλλοι ομιλητές. Θα ήθελα να είσαστε πιο συνεκτικοί από τους σκιώδεις. Σαρή Ισάια, Εσάια και μετά Τόμας Μάν. Ευχαριστώ θα χρησιμοποιήσω στη μητρική μου γιατί είναι δυνατό σε αυτή τη συνάντηση και ευχαριστώ τη Γραμματεία για αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το, την εισηγήτρια και τους σκιώδεις γιατί ξέρω ότι προέβησαν σε μια πολύμηνη εργασία για να φτάσουν σε μια κοινή θέση και είναι λυπηρό ότι στο παρελθόν ε, φτάσαμε σε, και τώρα φτάσαμε σε δύο σειρές ε, τροπολογιών συμβιβασμών που θα ψηφίσουμε αύριο. Αποστέλουμε ένα λανθασμένο μήνυμα νομίζω προς τα έξω, διότι αυτό που έχει σημασία είναι η βελτίωση της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην γίνει ε, υπεκφυγή και παράκαμψη των ρητρών της οδηγίας, ιδιαίτερα στα άρθρα 4, 5 και 6, 7 και 8 ως προς την ε, διοικητική συνεργασία. Ελπίζω ότι έστω και την ίστατη ώρα θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα συμβασμό. Μιλάμε για διοικητικές διαδικασίες. Δεν μπορεί να είναι και τόσο πια πολιτική υφή το θέμα. Όπως είπαν πολύ σωστά και οι σκιώδεις, τα 3, 9 ε, και 12 είναι τα τρία βασικά άρθρα. Το 3 αφορά την κατάχρηση και την παράκαμψη των διατάξεων. Θα πρέπει να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση στην απόσπαση των εργαζομένων, γι' αυτό και ο ανοιχτό κατάλογος είναι και ο μόνος ε, τρόπος ε, διεκπαιρέωσης, όπως είπε και η συγγήτρια. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή έθιξε ζητήματα όπως οι εταιρείες φραγίδες και την ανέντιμη εργασία που προτείνουν πολλοί ε, εργοδότες. Γι' αυτό επιβάλλονται οι εθνικοί έλεγχοι και να έχουμε έναν ανοιχτό κατάλογο έτσι ώστε ε, οι εθνικές διοικήσεις να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όσα μέτρα διαθέτουν για την απόσπαστη. Τα, μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα, ε, αναλογικά και να μην οδηγούν σε διακρίσεις. Η ερμήνεια αυτών των τριών λέξεων δημιούργησε πολλές αμφιβολίες και κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια ως προς την ερμηνεία έτσι ώστε να ε, μπορέσουν οι εθνικές κυβερνήσεις να δράσουν και να αντιμετήσουν τις, αντιμετωπίσουν τις εθνικές επιχειρήσεις σε σχέση με εκείνες των τρίτων χωρών. Δηλαδή δεν μπορούμε να θέτουμε απαιτήσει για επιχειρήσει ε, τρίτων χωρών τη στιγμή που δεν ισχύουν για τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά προβάλλουμε τον ε, προστατευτισμό και σε αυτή την περίπτωση η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ένα τιτάνιο έργο για να δει πού γίνονται οι διακρίσεις και πού όχι. Στο άρθρο 12 ο συμβασμός κάπως έχει αλλάξει, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα 27 κράτη-μέλη, σύντομα 28, αντιμετωπίζουν προβλήματα και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων που προβαίνουν στην απόσπαση. Γι' αυτό νομίζω ότι η εθνική ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Θα ήθελα να δούμε όλους τους μιλητές μαζί. Μασμάν ε, Υπάρχει κάποιος άλλος που ζητά το λόγο σε αυτή τη φάση, όχι. Τόμας Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καμιά φορά υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις. Όλοι από μας, όλοι μας μάλλον, επιθυμούμε να μας συγχαίρουν αλλά όλοι θέλουμε και την καθαρή γραμμή. Αύριο δεν έχουμε καθαρή γραμμή. Το είπαν διάφοροι συνάδελφοι. Πού οφείλεται αυτό. Αυτό οφείλεται και στο ότι ακόμα και μέσα στις πολιτικές ομάδες έχουμε αποκλίνουσες απόψεις. Να διασυμφωνώ συνήθως μαζί σου. Όταν μιλήσω όμως ότι υπάρχουν προσπάθειες προστατευτισμού, δεν το βλέπω αυτό. Εμείς θέλουμε να μπορεί να δουλεύουν λογικά, να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες εργασίας και στις χώρες αποστολής και στις χώρες υποδοχής των εργαζόμενων και γι' αυτό ευχαριστώ όλους τους κοιόδης εισηγητής. Μπόρεσα ξανά να μιλήσω με ορισμένους από εσά για να έχουμε μια συνολική προσέγγιση. Είπε η Ελίζα Μπετσουρέντερ ότι αύριο φοβάται ότι θα είναι χαόδηση η ψηφοφορία. Φοβούμαι ότι θα συμφωνήσω. Αγαπητή Περβάνς, μήπως υπάρχει κάποια δυνατότητα Μήπως υπάρχει κάποια δυνατότητα να πούμε ότι το αναβάλουμε. Αναβάλουμε την ψηφοφορία. Γιατί έχουμε τόσο αποκλίνουσες απόψεις, κάναμε κοινέ συνεντεύξεις τύπου, κάναμε από κοινού ε, προσπάθειες τροποποίησεων, έγιναν πολλές και σημαντικές διαπραγματεύσεις, αλλά δεν έχουμε κοινέ συμβαστικές τροπολογίε. Βλέπω ότι οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτες για το 3α προτείνουν οι χώρες μέλη να μπορούν να επιβάλλουν και άλλα επιπρόσθετα κριτήρια εφόσον δεν οδηγούν αυτά σε διακρίση. Εγώ συμφωνώ. Εν προκειμένου το ίδιο για την θέση που λέει όπως επιβεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές. Χαίρομαι που η Ντανούτα είπε ότι θέλουμε να ξεφύγουμε από τη δυνατότητα να λέμε notification και είπαμε πλέον information. Σημαντικό βήμα αυτό. Συμφωνώ και με την Elizabeth Βετσουέτερ, τον πράσινων, ναι, που λέει ότι notification για information, ναι, ανοιχτός κατάλογος, αλλά όταν λέει in advance, αυτό οδηγεί σε πλήρη αποδυνάμωση. Αυτό το βρίσκω και εγώ λάθος. Έχουμε πολύ διαφορετικές εμπειρίε εμπειρίες διάφορες χώρες μέλη και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να αποφευθούν αυτά τα λάθος μηνύματα. Δεν είναι δυνατόν έτσι εμφορούμενοι από ένα κοινό πνεύμα να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ λύσεις. Ίσως να παρακαθίσουμε όλοι σε ένα μεγαλύτερο κύκλο. Εμείς είπαμε από την αρχή να αποφύγουμε τις μαχητικές ψηφοφορίες εφόσον αυτό είναι, αυτό είναι δυνατό. Έχουμε καταφέρει να κινήσουμε πολλά. Για παράδειγμα στο άρθρο 12 όταν βλέπω εγώ την γερμανική διάταξη για την ε, συνολική, για τη γενική ευθύνη και αυτή τη λύση προτείνεται τώρα. Βρίσκω ότι είναι, ε, είναι ασημίβαστα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να έχουμε από την άλλη μεριά χώρες μέλη οι οποίες να μην θέλουν καμία λύση. Βλέπω προσπάθειες που γίνονται και από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Μήπως υπάρχουν και άλλοι. Καμιά φορά δεν είναι δυνατόν κάποιος να διστάζει ανάμεσα στη μια ή στην άλλη λύση. Ούτως ή άλλως το Σεπτέμβριο θα επανέλθουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε ένα περιθώριο ακόμα στους εαυτούς μας ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η ε, Περβάνος βλέπω ότι κάνει προχωρησουμε η σου βλεπω οτι κανει νευματα με το κεφάλι. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύγκριση αυτή των συμβαστικών τροπολογιών α ή β, της λίστας α ή της λίστας β. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή με θέτετε ενώπιον των ευθυνών μου για το θέμα αυτό, θα σας απαντήσω άμεσα και σας ευχαριστώ γιατί ως αντιπρόεδρος προσπαθήσατε να συνεισφέρετε έτσι ώστε είναι πιο αποδοτικές οι εργασίες μας. Θα ήθελα να επενθυμίσω στους συναδέλφους ότι όταν ε, βλέπουμε τις ε, αρμοδιότητες της Επιτροπής μας από την πρώτη μέρα της εκλογής ε, του Προέδρου Μπαρόζο, στη δεύτερη θητεία του, είχαμε δύο βασικά ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες μας. Το πρώτο ετέθη από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια ε, αναγκαία διαπραγμάτευση, αλλά ίσως υπερβολική των κοινωνικών εταίρων. Επρόκειτο για την οδηγία περί χρόνου εργασίας. Άρα θα λήξει αυτή η θητεία χωρίς οδηγία για το χρόνο εργασίας. Ο ε, κύριος Μπαρόζο εξελέγει με μια δέσμευση η οποία αμφισβητήθηκε από το σημείο εκκίνησης μετά από τις αποφάσεις Viking Λαβάλ και άλλων μετά από πιέσεις πολιτικών ομάδων για αναθεώρηση της οδηγίας. Άλλοι ήθελαν μια οδηγία ερμηνείας, καθαρά ερμηνευτική. Κατά τη στιγμή ανάληψης ε, της φοιτείας του Πρόεδρου Μπαρόζο, ο κύριος Μπαρόζο δεσμεύτηκε για την αναθεώρηση της ερμηνείας της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Η θητεία μας λύγει σε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο. Η συζήτηση μεταξύ σκιωδών που είναι αρκετά νεφελώδης, όπου δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη της Επιτροπής, αλλά μόνο η ομάδα διαπραγμάτευσης, είναι μια συζήτηση η οποία έχει αρχίσει εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν ξέρω πόσες φορές συνεδρίασαν οι σκιώδεις συνολικά, αλλά γνωρίζω ότι συνεδρίασαν αρκετές φορές. Και ο απόϊχος που είχα ήταν ότι δεν ήταν αποτελεσματικές αυτές οι συζητήσεις, γιατί αν κανείς ε, μετά από πολλοί μήνες συνεδριάσεις δεν φτάνει σε μία συμφωνία, σημαίνει ότι μιλάμε, πολλά, μιλάμε πολύ αλλά κάνουμε πολύ ο, λίγα. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές. Εγώ ξέρω την τακτική των διαπραγματεύσεων, ζητήματα τακτικής καθαρά. Και εγώ έχω πείρα στο θέμα, όπως και εσείς, και γνωρίζω ότι υπάρχει και η τακτική της καθυστέρησης που γνωρίζουμε πολύ καλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλω να μας κατηγορήσουν για την ίδια πρακτική. Και αν θέλουμε να έχουμε μία πιθανότητα να καταλήξουμε σε αυτό το κείμενο πριν από τη φοιτεία μας, θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Και μετά από αίτημα της εισηγήτριας της και της ομάδας μου ζήτησα την αναβολή. Τώρα τέλος, τέλος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και εσείς, και εσείς μου το ζητήσετε. Και η δική μου πολιτική ομάδα μου το ζήτησε. Δηλαδή αρκετές φορές ζητήθηκε αναβολή και πουθενά δεν είναι γραμμένο στον κανονισμό μας ότι πριν ψηφίσουμε στην ολομέλεια μιας επιτροπής θα πρέπει να υπάρχει συνένεση. Εάν υπάρχει διαφωνία, τότε θα ψηφίσουμε διαφωνώντας. Δεν θα ήθελα όμως να μην έχουμε θέση να μην ανοίξουν οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Και μη μου πείτε ότι χρειαζόμαστε άλλη μια μέρα. Όχι, τέλος, τέλος. Θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και θα ψηφίσουμε αύριο. Ε, Ρισάρ Φάμπρ και μετά Τσάμπα Όρη. a děláme, co děláme, postavení těch lidí, kteří budou vysíláni, se výrazně nezlepší. Ευχαριστώ. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα, πιστεύω, να είναι κανείς επιθετικός. Εδώ από ό,τι φαίνεται, η συγκίτρια μάλλον είναι κατά οποιασδήποτε πρόταση έρχεται από τους σοσιαλιστές ή από τα συνδικάτα. Αν δεν υπήρχαν οι σοσιαλιστές και τα συνδικάτα, δεν θα υπήρχε ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, αυτό, το οποίο, αυτό στο οποίο όλοι επιτίθενται σήμερα. Μπορεί κανείς να διαφωνεί, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να βγάλουμε από εδώ οποιαδήποτε πρόταση των σοσιαλιστών λέγοντας ότι δεν έχει νόημα. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για την προστασία από το κοινωνικό ντάμπινγκ. Έρχομαι εγώ από μια χώρα, την Τσεχία, όπου επικρατεί μαφιόζικος καπιταλισμός. Και νομίζω ότι και σε άλλες χώρες μετά την κομμουνιστική περίοδο το ίδιο ισχύει. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λένε ότι τα σουηδικά συνδικάτα δεν λειτουργήσαν καλά με τις θέσεις που αποφάσισαν σε σχέση με τους αποσπασμένους υπαλλήλους, εργαζόμενους. Πρόκειται πάντα για διεθνείς οργανισμούς που προσπαθούν να δουν κατά πόσο τα συνδικάτα συμπεριφέρθηκαν όπως έπρεπε ή όχι, τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν τα συνδικάτα. Οπότε τελικά τα συνδικάτα φοβούνται. Στις παλιές χώρες μέλη υπάρχει ήδη ένα επίπεδο προστασίας. Δεν μπορεί κάποιοι που μεταφέρονται και πηγαίνουν κάπου αλλού να ζουν κάτω από χειρότερες συνθήκες και ούτε μπορούμε τώρα να προσπαθούμε να αλλάξουμε όλες τις συνθήκες. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα, χωρίς να επιτιθέμεθα ένα στον άλλον η οδηγία που υπάρχει δεν είναι σαφής. Κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Στην Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε αποτελέσματα, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι σε όλες τις χώρες μέλη να μπορούν να επωφεληθούν και να αποφύγουμε να τα βάζουμε με την επικουρικότητα, να μιλάμε για αυτήν ή για άλλα ούτε ανοιχτό συντονισμό. Όλα αυτά είναι ψευδέστηση. Τσίβι, Και ποιο άλλο θέλει το λόγο, ή να κλείσω τον κατάλογο. Ο Μίλητον, και εγώ θέλω να πω δύο λόγια μετά. Εντάξει, ωραία. Παρακαλώ, κύριε Ορί. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα ήδη υπόθηκαν. Έχω όμως και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. θεωρώ ότι δεν υπάρχει τρόπος να δακτυλοδειχτούμε ο ένας τον άλλον. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι πράγματι οι θέσεις μεταξύ μας είναι πολύ μακριά. Και όχι μόνο μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αλλά όπως είπε και ο Τόμας Μαν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποια γλώσσα με τη διερμηνία. Τώρα είναι εντάξει. Συνεχίζω λοιπόν, ή μάλλον ξαναρχίζω, λέει ο μιλητής. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να δακτυλοδεικτούμε ένα τον άλλον. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις, υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου διαφαίνονται βασικές διαφορές. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και τώρα. Επιπλέον, οι διαφορές αυτές δεν είναι πάντα μεταξύ πολιτικών ομάδων, μερικές φορές είναι και μέσα στην ίδια την πολιτική ομάδα ή μεταξύ των ε, μελών που προέρχονται από την ίδια χώρα. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για διαμάχη εδώ Ανατολής Δύσης. Αν δούμε τι γίνεται με την κοινωτικότητα των αποσπασμένων εργαζόμενων, έχουμε πολύ περισσότερους αποσπασμένους εργαζόμενους από τις ε, παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά από τις καινούργιες. Άρα αν υπάρχει κίνδυνος για κοινωνικό ντάμπινγκ δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί μεγαλύτερος. Η δουλειά που έκανε η Ντανούτα μέχρι τώρα πιστεύω ότι είναι αξιοπρόσεκτη. Προσπάθησε τα πάντα για να προσεγγίσει θέσεις οι οποίες αρχικά ήταν πολύ μακριά μεταξύ τους και για να πετύχει σε βιβασμούς η ίδια η πρόεδρος είπε ότι η θέση δεν είναι σαφής. Ναι, μα ακριβώς προσπαθώντας να πετύχει σε βιβασμούς, οδηγήθηκε εκεί η συγκήτρια στην αρχή. Η θέση της ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αν τώρα είναι λιγότερο συγκεκριμένη είναι γιατί προσπάθησε να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις και γιατί έδειξε τεράστια καλή θέληση για να προσεγγίσει τις διαφορετικές απόψεις. Γι' αυτό και σήμερα η θέση της ίσως να μην είναι τόσο σαφής. Ακόμα και αν αρνήθηκε πρόεδρος την ιδέα, εγώ δεν νομίζω ότι είναι πραγματικά αδύνατο να ακολουθήσουμε την πρόταση του Τόμας Μαν. Καταρχήν, συμφωνώ για το ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την άποψη του Συμβουλίου. Μπορούμε να διατυπώσουμε τη δικιά μας άποψη. Αλλά αφού ξέρουμε ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια κατάσταση όπου έγινε με το Ταμείο για τους Άπορους όπου είμαστε εμείς έτοιμοι και δεν είναι το Συμβούλιο. Εξάλλου ξέρουμε ότι αυτή τη εβδομάδα στην ε, συνάντηση που έγινε θα υπάρξει μια έκθεση πρόοδου επί της ουσίας για την απόσπαση. Λοιπόν, μπορούμε να είμαστε έτοιμοι μέχρι τέλη Ιουνίου ή Ιουλίου, αλλά να είμαστε εμεί έτοιμοι και να μην είναι το Συμβούλιο. Δεν λέω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τη θέση του Συμβουλίου, αλλά λέω ότι καλό είναι να λάβουμε υπόψη μα ποιο είναι το πλαίσιο και να είμαστε ρεαλιστέ. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε. Πάντω, όντω είναι τα άρθρα 3, 9 και 12 εκείνα ε, τα οποία δημιούργησαν τις περισσότερες συζητήσεις και διαφωνίες, πολιτικές συζητήσεις και μάλιστα πολλές φορές με μεγάλη αίσθηση. Και αυτό πιστεύω εξαιτία της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες μέλη. Δεν καταλήξαμε σε μια καλή λύση. Δεδομένης της νομοθεσίας, η νομοθεσία πάντα βρίσκεται πίσω. Αν το μελετήσετε το θέμα θα δείτε ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αν αρνηθούμε πλήρως να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη φύση της νομοθεσίας, ότι πάντα είναι πιο πίσω, θα δημιουργηθεί αναρχία. Γιατί ο νόμος καθορίζει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Και όταν ο νόμος αυτός διαφέρει από την πραγματικότητα, τότε πρέπει να αλλάξει. Εδώ αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 9. Προκειμένου κάποιος, για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε, να μπορεί να βάζει εμπόδια στην απόσπαση των εργαζομένων, πολλέ τροπολογίε πάνε, θυμίζω, προ αυτή την κατεύθυνση, αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε, ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να δημιουργήσει τέτοια εμπόδια. Ε, εγώ διαφωνώ. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι νομική ασφάλεια και δεν μου κάνει εντύπωση που προσπαθεί να βρει σε βιβασμού η Ντανούτα, αλλά δεν μπορεί να φτάσει και μέχρι εδώ, γιατί πρόκειται για υπερβολές. Δεν συμφωνώ και με τον ε, Ρίτσαρτ, ακόμα και αν ε, σέβομαι την άποψή του. Δεν, ότι δεν δέχτηκε καμία πρόταση των συνδικάτων η Ντανούτα, δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ιδέα που λέει ότι τα συνδικάτα μπορούν να έχουν την ίδια εντολή που έχουν και οι αρμόδιες αρχές γιατί τότε πρόκειται για έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους και πρόκειται για συνεργασία ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Καμία από τις δύο πλευρές δεν πρέπει να βρεθεί σε τέτοια κατάσταση που να έχει τις ίδιες αρχές τι ίδιε συγγνώμη αρμοδιότητε όπω έχει η ελεγκτική αρχή. Η ελεγκτική αρχή υπάρχει γιατί ακριβώ πρέπει να είναι ανεξάρτητη ούτε με του μεν ούτε με του δε. Και πρέπει να γίνεται σεβαστή η άποψή τη στα νομικά κείμενα και νόμοι. Εδώ υπάρχει υπερβολή λοιπόν. Είναι επίσης λυπηρό που πρέπει τώρα να βρούμε προτάσεις ανάμεσα σε αυτά τα δύο πακέτα συμβασμών. Αν η Πρόεδρος θεωρεί ότι είναι πολύ μακριά οι θέση των ΜΕΝ και των ΔΕ και άρα δεν μπορούμε να καταλήξουμε πουθενά, ναι, όντως η λίστα μπορούσε να ήταν να ψηφίσουμε και θα δούμε. Αυτοί όμως που λένε ότι υπάρχει προσέγγιση αλλά δεν έχουμε πετύχει αρκετή προσέγγιση, τότε εκείνοι έχουν δίκιο που λένε ότι πρέπει να έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας για να πετύχουμε την πλήρη αυτή προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ πάντως ε, την εισηγήτρια. Η Πρόεδρος αναφέρθηκε και σε κάτι ακόμα. Η οδηγία για το χρόνο εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι δεν φταίει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν προχωρήσαμε το Κοινοβούλιο είχε μια συνεπή θέση, αλλά όχι ελαστική για το opt-out, για παράδειγμα. Η συνέπεια είναι ότι η... φάνηκε ότι πηγαίναμε πέρα από τις νομικές μας αρμοδιότητες και η συνέπεια είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε ακόμα πιο μακριά από την επιτευξή συμβιβασμού από ό,τι βρισκόμασταν πριν από πέντε χρόνια. Θα ήταν καλό λοιπόν τώρα για την απόσπαση να αποφύγουμε μια αντίστοιχη κατάσταση και να μην βρεθούμε τελικά ακόμα μακριά από το σημείο εκκίνησης και δεν ε, μπορούν να γίνουν ε, σεβαστά και να προστατεύονται τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζόμενων. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε. ο κύριο Σέρκας. Τέθηκε το θέμα να ψηφίσουμε ή να μην ψηφίσουμε σήμερα. Το είπε και ο κύριος Όρη. Εγώ θέλω να σας πω ποια είναι η άποψη των σοσιαλιστών. Πολλέ φορέ ζητήσαμε από την Πρόεδρο να αναβάλει την ψηφοφορία για να επιτευχθεί συμφωνία. Και δεν αποδείχθηκε εφικτό. Είναι τελευταία ευκαιρία που έχουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας. Να, τη... να σεβαστούμε τους εαυτούς μας και να μας σεβαστεί και το Συμβούλιο. Γι' αυτό προτείνουμε να ψηφίσουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν μπορούμε να μπούμε και να κάνουμε το ίδιο που κάνει και η Επιτροπή, να καθυστερεί. Όχι. Το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφανθεί και η Δημοκρατία αυτό θέλει. Όποιος ε, κερδίσει, κέρδισε. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά να κάνω μερικές παρατηρήσεις επί της ουσίας. Η πρώτη μου παρατήρηση έχει να κάνει με το τι διακυδεύεται με την οδηγία αυτή. Ο Θαβαωρή είπε ότι δεν θέλουμε να βάλουμε εμπόδια στην απόσπαση των εργαζομένων. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιο είναι το αντικείμενο της οδηγίας αυτής. Είναι να επιτρέπεται η προσωρινή απόσπαση για την παροχή μιας υπηρεσίας. Αν αναθεωρούμε σήμερα την οδηγία αυτή είναι γιατί διαπιστώσαμε ότι για αυτή την προσωρινή απόσπαση για την παροχή μια υπηρεσίας του εργαζόμενου οδηγηθήκαμε σε κατάχρηση της οδηγίας αυτής και διαπιστώσαμε ότι τελικά αποσπώνται οι ΣΕΗ, οι εργαζόμενοι, κάτι το οποίο αποσταθεροποιεί την αγορά εργασίας της χώρας προέλευσης των εργαζομένων αυτών. Λαμβάνοντα υπόψη μα ε, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, λέμε ότι αυτό γίνεται πιο ευάλωτο, πιο εύθραυστο. Ω Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνε μας, πιστεύω, για αυτό ακριβώ το οποίο διακυδεύεται με την οδηγία αυτή και για τις συνέπειες που έχει όχι μόνο στον κοινωνικό τομέα αλλά και στον πολιτικό. Για την ψηφοφορία. Θα λάβει χώρα αύριο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 24 ώρες στη διάθεσή μας. Όσοι θέλουν να βοηθήσουν στην προσέγγιση των απόψεων μπορούν. Η ψηφοφορία όμως θα λάβει χώρα αύριο. Για το αν πρέπει ή όχι να περιμένουμε το Συμβούλιο τώρα. Το έχω ήδη πει ότι όλα είναι δυνατά. Υπάρχουν καταστάσεις όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει μετά το Συμβούλιο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Κοινοβούλιο ψηφίζει πριν από το Συμβούλιο. Το κάθε θεσμικό όργανο δρά αυτόνομα, με το δικό του ρυθμό. Ο ρυθμός ο δικός μας ήταν ένας σοβαρός ρυθμός, με συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών, και από ό,τι άκουσα από αυτά που είπατε, οι συνεδριάσεις αυτές ήταν πυκνές, κρατούσαν πολλή ώρα, τα επιχειρήματα ήταν πολλά που ακουγόντουσαν εκεί, οπότε το ότι πάμε γρήγορα, βιαζόμαστε και μετά θα πρέπει να καθίσουμε και να περιμένουμε το Συμβούλιο, δεν στέκει γιατί είμαστε αυτόνομο όργανο. Έπειτα άκουσα την εισηγήτρια να λέει. Και εδώ βέβαια δεν μιλάω ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Ως μέλος της Σοσιαλιστικής Ομάδας μιλάω. Σας άκουσα αγαπητή συγκίτρια να λέτε ότι οι σοσιαλιστές πρότειναν την ελεύθερη εκπροσώπηση των εργαζομένων χωρίς τη δικιά τους τη συνένεση. Ξέρετε, πήγα κι εγώ και με άλλους στη Φλαμανδίλη και είδα ποια είναι η κατάσταση των Πολωνών εργαζόμενων εκεί, οι οποίοι είχαν ένα συμβόλαιο στα αγγλικά μια ολόκληρη σελίδα που δεν μπορούσαν καν να διαβάσουν και να καταλάβουν. Καμία εκπροσώπηση. Είδε επίσης τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εκπροσωπούνταν και πόσο ευτυχής ήταν αν υπήρχε μια μικρή μία, μικρή μη κυβερνητική οργάνωση με έναν να μιλάει λίγα πολωνικά για να μπορεί να τους ακούσει. Στο χαρτί με το μισθό τους έλεγε τι έπρεπε κανονικά να τους κρατάνε για φόρους, ασφάλιση κτλ. Τίποτα δεν υπήρχε που να καταλαβαίνουν. Για μένα λοιπόν η διατύπωση η οποία περιλαμβάνεται στο συμβασμό των σοσιαλιστών είναι τεράστια σημασίας. Γιατί όλοι συμφωνούμε με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το συνδικαλιστικό δικαίωμα, για την εκπροσώπηση των εργαζομένων, αλλά όλα αυτά πούντα πρέπει να υπάρχει πραγματικό δικαίωμα των εργαζομένων. Και αν θέλουμε πραγματική εκπροσώπηση των εργαζομένων, τότε πρέπει να ακολουθήσουμε την τροπολογία αυτή των σοσιαλιστών. Δεύτερον, επί της ουσίας, υπάρχει κάτι που με θλίβει και το λέω και στις δυο ομάδες, γιατί η κοινή και αλληλέγγυα ευθύνη δεν υπάρχει πια. Και αυτό με λυπεί αφάνταστα. Γιατί στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό. Και διαπιστώνω ότι με τις διαπραγματεύσεις και με την τέχνη αυτή του συμβιβασμού χάσαμε. Αυτό το οποίο σημαίνει κάτι σημαντικό όσον αφορά τα δικαιώματα και κάτι που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Το λέω αυτό σε όλους ότι λυπάμαι πολύ που δεν υπάρχει πια στο κείμενο. Τέλος. αλλά το λέω κάπως στο περιθώριο, γιατί βέβαια τα ουσιώδη έχουν συζητηθεί. Είναι το γλωσσικό, το θέμα των γλώσσων. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νάντια Χίρς, με εκπλήσει. Έρχεστε από μια χώρα η οποία καθημερινά ζητάει η δικιά σας η γλώσσα να λαμβάνετε υπόψη παντού και κάθε φορά που χρειάζεται δέχεστε ένα συμβιβασμό σύμφωνα με τον οποίο οι εργοδότες οφείλουν μόνο στα αγγλικά να παρουσιάζουν τα έγγραφά τους. Μα οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι είναι αποσπασμένοι στον οικοδομικό τομέα, στις μεταφορές ή και στη γεωργία. Η εργοδοσία στους τομείς αυτούς πολύ συχνά αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν ξέρουν καθόλου αγγλικά. Να μιλάμε λοιπόν από το σύνολο των εργαζομένων και από το σύνολο της εργοδοσίας. Επειδή θέλουμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη των εργαζομένων, να τους υποχρεώσουμε όλους να μιλάνε αγγλικά, δεν θεωρώ ότι είναι αποδεκτό. Κοιτάξτε το συμβιβασμό που προτείνει η συγκήτρια και θα καταλάβετε τι εννοώ. Συγγνώμη που υπογράμμισα αυτές τις λεπτομέρειες αλλά μια που δεν είχαν αναφερθεί από τους υπόλοιπους, γι' αυτό τα λέω. Τώρα, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως σύντομα θα μπορούσε... Α, δεν θέλει να παρέμβει. Κατάλαβε. Μην εκνευρίζεστε, κυρία Συγήτρια. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Θα σας δώσω το λόγο, χωρίς καν να τον έχετε ζητήσει, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Προηγουμένως, σας λέω ότι έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας αν θέλουμε να τηρήσουμε το ωράριό μας, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι καθόλου θυμωμένη, δεν έχω εκνευριστεί καθόλου. Απλώς ήθελα να λάβω θέση σε σχέση με τις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν, γιατί η παρούσα κατάσταση δεν είναι απόλυτα ε, σαφής. Γι' αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα πριν από την αυριανή ψηφοφορία. Σε σχέση με τον Στίβεν Χιούς. Στίβεν, Μίλησες για μία ε, δημόσια οριοθέτηση. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν ε, πολλές δυνατότητες εφαρμογής του προστατευτισμού. Γι' αυτό εμείς αντιταχθήκαμε σε αυτή την οριοθέτηση. Μίλησες για την αναλογικότητα και για το βάσιμο της πρότησης. Αυτή είναι βασική όρη ε, σύστασης οποιασδήποτε νομοθεσίας. Θέλουμε να εξαλείψουμε τις εταιρείες ε, σφραγίδα, καταρχήν. Και μιλάμε για αναλογικότητα γιατί θέλουμε να ξέρουμε αν κάτι είναι νόμιμο ή μη. Σας έδωσα το παράδειγμα του, του μεγέθους του παπουτσιού. Για να υπάρχει ισότητα θα πρέπει ο νόμος να ισχύει για τους ντόπιου και μη ντόπιου. Να ισχύει η ίδια νομοθεσία. Στίβεν, θα πρέπει να μιλήσουμε και να προβάλλουμε τις απόψεις μας μέσω μίας και ενίας ιστοσελίδας. Έδωσε στο παράδειγμα της Γερμανίας. Δεν πρόκειται για μία ενιαία πηγή πληροφόρησης, πρόκειται για μία ιστοσελίδα, για μία διαδικτυακή πύλη. Εκεί θα υπάρχει ενιαίος χαρακτήρας για να υπάρχει και νομική ασφάλεια. Και επιπροσθέτως πέρα δηλαδή από την ενιαία αυτή πηγή πληροφοριών θα έχουμε τη δυνατότητα συμπλήρωσης με άλλες πληροφορίες γνωρίζοντας ότι πάντα υπάρχουν επιφυλάξεις και μπορούμε να έχουμε και επιπρόσθετες πηγές και καλύτερα διαρθρωμένες. Σε σχέση με τις αρμόδιες αρχές, Υπάρχει μεγάλο χάος στους σοσιαλιστές που θέλουν να επιβάλλουν ένα πρότυπο επιθεώρησης εργασίας και θέλουν να επιβάλλουν τη θέση τους στα συνδικάτα. Άρα τα συνδικάτα θα λάμβαναν όλες τις διοικητικές πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια τα συνδικάτα θα μπορούσαν να ζητήσουν ελέγχους και κυρώσεις στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι χαόδες. Νομίζω ότι κάθε εθνική ε, διοίκηση είναι αρκετά αποτελεσματική για να επιβάλλει αυτές τις υποχρεώσεις. Ποιος θα χρηματοδοτούσε εξάλλου κάτι τέτοιο. Είπες ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα των κατασκευών υποστηρίζουν τις προτάσεις των σοσιαλιστών. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις που υποστηρίζονται και από τους εργοδότες. Γιατί πολύ συχνά προβάλλεται τις απόψεις σας που λαμβάνω και εγώ με τη σειρά μου Υπάρχει όμως μια πληθώρα θέσεων που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, που προέρχονται όλες από τους σοσιαλιστές. Ε, ποιες ε, θα υποστηρίξουμε. Νάντια Χίρ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το άνοιγμα που δείχνεις ε, και που η ομάδα σου άνοιξε τα χαρτιά της, διότι ήταν η πιο ανοιχτή ομάδα στις προτάσεις και από, τη δική μας πλευρά και των σοσιαλιστών και των πρασίνων. Συμφωνώ μαζί σου ότι για να μπορέσουν οι εργοδότες να προστατεύσουν τους εργαζόμενους θα πρέπει να προστατεύονται και οι ίδιοι. Ελίζαμπετ, έχεις δίκιο. Η νομοθεσία θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και ε, διαρκή στο χρόνο. Η εργασία της ομάδας σου ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη. Είπες ότι η ψηφοφορία θα είναι χαοτική. Δεν ισχύει αυτό εάν είμαστε πραγματικά υπεύθυνοι για τους εργαζόμενους, υπέρ των εργαζομένων, ξέρουμε πώς να ψηφίσουμε. Τόμας Χέντελ επέσυρε την προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχουν ε, ορισμένα, ορισμένα σφάλματα της ε, γραμματείας σε σχέση με το άρθρο 19. Ε, Ζήτησα από τη γραμματεία να το επαληθεύσει. Richard θα ήθελα να απαντήσω λέγοντας ότι ίσως ήμουν ιδιαίτερα ζωηρή στις αντιδράσεις μου, αλλά ξέρω πολύ καλά τι συνέβη. Ήταν πολύ οι διαπραγματεύσεις και δεν σύμφωνο με την ε, πρόεδρο που είπε ότι δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί και εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια όπου κατά τη δεκαετία του 90 είχαμε πολλούς αποσπασμένους και από το 96 συνεργάζομαι με τις ε, ε, οργανώσεις των εργοδοτών για τους αποσπασμένους δεν αντιτίθεμε στην εργασία των αποσπασμένων. Τα συνδικάτα ε, με απείλησαν με απεριακές κινητοποίησεις. Τώρα όμως θα ήθελα τα συνδικάτα να οργανώσουν απεργίες στην περιφέρειά μου, διότι μπορώ να τους επεξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα και πόσο έχω εργαστεί για τους αποσπασμένους. Τέλος, θα ήθελα να απαντήσω στην Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ως προς τον ρόλο των συνδικάτων. Τα συνδικάτα θα πρέπει να ανησυχούν για το μέλλον των εργαζομένων. Είναι δύσκολο να αντιτασσόμαστε πάντα στους εργοδότες και τα συνδικάτα ε, ανταποκρίνονται πολύ καλά στο ρόλο τους. Μην ξεπερνάμε όμως τις κόκκινες γραμμές ε, αποδίδοντας τα συνδικάτα ένα ρόλο που δεν έχουν. Δεν μπορούν να ε, προβούν στην αντικατάσταση ή στην υποκατάσταση των εργαζομένων. Νομίζω ότι τότε ξεπερνάμε ένα νομικό στάτους κβό, κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει. Αυτό το σχέδιο έκθεσης καταρτίστηκε όχι μόνο από την υποφαινόμενη και τους σκιώδεις και από τη γραμματεία, αλλά και από δεκάδες μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας τροφοδότησαν με τη θέση τους. Και επειδή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας είχαμε συνεχείς επαφές με τις πολιτικές μας ομάδες, γι' αυτό ε, χρειάστηκε να χρονοτριβήσουμε κάπως. Ήταν δηλαδή κάπως χινοτενής η διαδικασία. Δεν πρόκειται μόνο για τους αποσπασμένους και για την οδηγία, για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και την κρίση. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε, βρισκόμαστε στο ίδιο ηλικιακό φάσμα και καταλαβαίνουμε ορισμένα πράγματα. Δεν μιλάμε για την απαρχή και για την αρχή και το τέλος της εργασίας. Βρισκα, βρισκόμαστε στην ε, σε μια συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση και συμφραζόμενα έχουν αλλάξει οι καιροί και θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να βρούμε τη σωστή μας θέση κάτω από τον ήλιο. Εάν αύριο υπερψηφίσουμε τη θέση των σοσιαλιστών, τότε θα αποτύχω εγώ. Ε, δεν θα ε, υπερασπιστώ τους αποσπασμένους. Ένα εκατομμύριο αποσπασμένοι θα χάσουν τη θέση εργασία τους και έτσι θα αυξήσουμε και το δίκτυο ανεργίας τις σειρές των ανέργων, κάτι το οποίο δεν επιθυμεί η ευρωπαϊκή κοινωνία αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ωραία, η Πρόεδρος. Τελειώσαμε με την γενική συζήτηση και θα τα πούμε σήμερα το απόγευμα για τη συνέχεια των εργασιών μας ε, ε, για την έκθεση της κυρίας Ντανούτα Χούμπνερ. Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί ε, αύριο. Με, με συγχωρείτε ενό την έκθεση της Ντανούτα Γιατσλοβίτσκα η οποία θα ψηφιστεί αύριο το πρωί όπως προβλεπόταν αρχικά.